Αγαπητοί συνάδελφοι. Άρχεται η συνεδρίαση, αρχίζουμε τις εργασίες μας. Ε, παρακαλώ ε, ησυχία. Είναι σημαντική η συνάντησή μας σήμερα και αύριο. Έχουμε σημαντικές ψηφοφορίες. Θα αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, θα ήθελα... Παρακαλώ ησυχία. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω στους συντονιστές ότι επειδή πήγε καλά η συνεδρίασή μας σήμερα το πρωί, δεν χρειάζεται να ξαναβρεθούμε στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ωραία. Για την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Σας προτείνω να περάσουμε στην ψηφοφορία για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση να ψηφίσουμε τις μεταφορές πιστώσεων για ε, το Ταμείο αυτό αμέσως μετά τις ε, ε, εν λόγω ενέργειες. Όσον αφορά τις αναγγελίες του Προέδρου, υπάρχουν ήδη στα κείμενά σας άλλες ε, παρατηρήσεις, ανακοινώσεις, συγγνώμη, ενημερώθηκα ότι στο σημείο 14 του ενημερωτικού κειμένου που έχετε λάβει υπάρχει ένα πρόβλημα με τα στοιχεία. Αντί για 4.300.000 κτλ. είναι 2,29 κλπ. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης μας 19 Σεπτεμβρίου. Παρατηρήσεις. Όχι. Θεωρούμε, θα θεωρήσουμε ότι ενεκρίθησαν στο τέλος της συνεδριασής μας αν δεν έχουν υπάρξει παρατηρήσεις και περνάμε απευθείας στον προπολογισμό 2013. Σας προτείνω, επειδή η Φραντσέσκα είναι στην ώρα της, να ψηφίσουμε ίσως πρώτα το σχέδιο διορθωτικού προπολισμού το σημείο 4. Έλγα, ευχαριστώ. Θα πρότεινα να ψηφίσουμε για το EDF σήμερα το απόγευμα. Γιατί δεν έχουμε ακόμη για το EGF μάλλον, το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση σήμερα το απόγευμα. Α, για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μόνο. Υπάρχουν αντιρρήσει. Η κυρία Τρίπελ, θέλουμε να καταλήξει ο κατάλογος προφοριών. Δεν υπάρχει πολιτικό πρόβλημα. Θέλουμε απλώς ε, να είναι πιο λειτουργική η ψηφοφορία. Έτσι είχε προγραμματιστεί, συνεχίζει η κυρία Τρίπελ. Πρόεδρος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν δεν υπάρχει πρόβλημα για κανέναν, θα ψηφίσουμε για το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση το απόγευμα. Σας προτείνω λοιπόν να αρχίσουμε με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθμός 4. Η Φραντσέσκα και μετά θα περάσουμε στον προϋπολογισμό του 13. Φραντσέσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήδη συζητήθηκε το έγγραφο αυτό δύο εβδομάδες πριν. Είναι ένα έγγραφο με πολλά τεχνικά σημεία. Μετά τις συζητήσεις αυτές προτείνω να υπερψηφίσουμε. Υπέρ και των δύο τροπολογιών Γκρέσλε και την ευχαριστώ γιατί οπωσδήποτε βελτιώνουν το κείμενο. Ευχαριστώ. Très bien. On peut voter en bloc. Ωραία, να τις ψηφίσουμε από κοινού και τις δύο. Ποιοι είναι υπέρ των δύο τροπολογιών. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Ομόφωνα. Για άλλη μια φορά θρίαμβος της ε, κυρίας Ίνιε Γκρέσλε. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροποποιημένη λοιπόν τώρα έκθεση σας προτείνω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε ότι λειτουργεί ε, το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορία, ότι ο Σαλβαδόρ έχει την κάρτα του και ότι δεν έχει υπερβολικά πολλούς του ΕΛΚΑ στην αίθουσα. Τελική λοιπόν ψηφοφορία. Α, ούτε η Ίγκε έχει κάρτα, αλλά έχει δικαίωμα ψήφου. Ούτε ο Σαλβαδόρ. Και η Αγγέλικα Βέρτμαν χρήσιμο βλέπετε να κάνουμε ψηφοφορίες. Μόνο 30 συνάδελφοι έχουν τις κάρτες τους και ψηφίσατε μόνο 28. Ωραία. Φέρανε βοηθή του Σαλβαδόρ την κάρτα του. Πέρασε. 27 υπέρ, 28. 0 κατά, τρεις αποχές. Εντάξει. Συγχαίρουμε λοιπόν την Φραντσέσκα. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 4 ψηφοφορία επί του κοινού ψηφίσματος των δύο εισηγητών μας για τον προϋπολογισμό του 13. Θέλουν το λόγο οι εισηγητές. Τζοβάνι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν πρόκειται για δήλωση, απλώς μία εισαγωγή στην ψηφοφορία κατά κάποιο τρόπο, γιατί σημείο εκκίνησης είναι η ανάκτηση δύο θεμάτων που ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα που όμως θα πρέπει να προσαρμοστούν κάπως. Πρόκειται για τεχνική προσαρμογή για να συμβαδίσουμε με τις συμφωνίες με τους συντονιστές. Γιατί τα καταφέραμε μεν στην ψηφοφορία, αλλά δεν πήραμε όλες τις σκόπιμες αποφάσεις. Το πρώτο θέμα αφορά τις, τους οργανισμούς οικονομικής εποπτείας με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού της Κομισιόν και για λόγους συνέπειες, συνέπειας, για να μην αυξηθούν τα διοικητικά έξοδα, έχουμε μία προσαρμογή. Έχουμε προσαρμόσει τα ποσά για να ακολουθήσουμε την Επιτροπή ΕΚΟΝ, τις τροπολογίες της. Για τους τρεις οργανισμούς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη θετική ψήφο της ΕΚΟΝ. Η δεύτερη προσαρμογή αφορά μία τροπολογία της ΙΜΚΟ που θέτει σε αποθεματικό 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η αρχική πρόταση της ΙΜΚΟ μιλούσε, έκανε λόγο για 2,3 εκατομμύρια. Άρα, στο αποθεματικό Στη γραμμή 120201 βάζουμε μόνο 1,5 εκατομμύριο. Αυτό το συμφωνήσαμε σήμερα το πρωί και με τους συντονιστές και υπήρξε ευρύτατη συμφωνία ως προς τη γραμμή αυτή. Δεύτερον, μία προφορική τροπολογία που θα πρέπει να ψηφίσουμε πριν αρχίσουμε με την ψηφοφορία καθεαυτή που αφορά την πρώτη προφορική τροπολογία που βλέπετε στον κατάλογό σας. που αφορά το εξή θέμα. Το ότι δεν λαμβάνουμε όλες τις γνωμοδοτήσεις των εξειδικευμένων επιτροπών. Δεν θα τις ψηφίσουμε λοιπόν, γιατί είχαμε πολύ περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας. Έχουμε την προφορική στην αιτιολογική σκέψη α που βρίσκεται σε σελίδα 13 του καταλόγου. Σελίδα 13. Ευχαριστούμε Τζοβάνι. Ντέρεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εντάχει. Ό,τι αναλαμβάνουμε, όταν γίνεται η ψηφοφορία, κοιτάμε τον εισηγητή για να δούμε αν αντιτίθεται ή όχι. Στο 1, στην 1.29 δεν θα κάνω υποδείξεις και προτείνω ε, καταβούληση ψήφο στην 129. Γιατί φτάσαμε στην τροπολογία συμβιβασμού 6 που καλύπτει πολλά θέματα και επί της ουσίας λέει ότι θα πρέπει να αναπέμψουμε όλα αυτά τα θέματα στις ε, εμπλεκόμενες επιτροπές. Επίσης υπάρχουν και δύο τεχνικές, ε, ψηφο, τεχνικής φύσης ψηφοφορίες, ε, μάλλον τροπολογίες, οι οποίες δεν, δεν αναφέρονται στον κατάλογο ψηφοριών. Χαρτόγκ. Στην 6, στην τροπολογία συμβασμού 6, και ως προς αυτήν θεωρώ ότι η 136 την καλύπτει. Θα ήθελα να γίνει ξεχωριστή ψηφοφορία, διότι δεν είμαι και ιδιαίτερα υπέρμαχος αυτής. Ωραία. Θα λάβουμε υπόψη αυτή την θετική σας σκέψη. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Πρώτο, θέμα ως προς τις ε, τεχνικές διορθώσεις του Τζοβάνι Λαβία που εντάσσονται σε έναν πίνακα που έχετε μπροστά σας. Υπέρ παρακαλώ, του πίνακα αυτού. Κατά. Ένας κατά. Δύο αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν ο πίνακας. Περνάμε τώρα στον κατάλογο ψηφοφοριών με την προφορική τροπολογία που υπέβαλε ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Ένας κατά. Αποχές. Δύο αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. Ένα, Φερέιρα. Ο εισηγητής ε, τίθεται κατά υπέρ παρακαλώ η Γκουε κατά. Πολλοί άλλοι αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 1. 2. Των σοσιαλιστών και δημοκρατών ο εισηγητής έχει τεθεί κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 της Γκουε. Εισηγητής κατά. Υπέρ παρακαλώ. 3. Κατά. Η πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται κατά σύνεπη. Τροπολογία 4. Έλγα ΤΡΟΥΠΕΛ. Ο εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ. Κατά. Τρεις αποχές. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια έχουμε τέσσερις ε, ψηφοφορίες του κυρίου Φεϊραήρα. Ο εισηγητής είναι κατά. Μπορούμε να τι ψηφίσουμε από κοινού. Υπέρ των τεσσάρων. Ουδής, ουδής. Κατά. Αποχές. Ωραία, απορρίπτεται. Κατά συνέπεια, κανείς δεν είναι υπέρ. Έχουμε δύο συμβατές τροπολογίες. Την 9 Ashworth, ο εισήτης είναι κατά, υπέρ παρακαλώ. Ένας, κατά. Η πλειοψηφία, αποχές, απορρίπτεται. δέκα. Φέρμ, καρδιά θα πάλι, πέρ. Ο εισηγητής είναι κατά. Οι σοσιαλιστές. Και η Γκουε. Ψηφίζουμε την 10. 10. Η Γκουε και οι σοσιαλιστές είναι υπέρ, κατά. Όλοι οι άλλοι κατά, αποχές, άρα απορρίπτεται. Συμβιβασμός 1, επί της παραγράφου 3. Υπέρ παρακαλώ, κατά, 9. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα, περνάμε στην 15 της Helga Truppel που είναι συμβατή. Γιατί μιλάμε για εισαγωγή νέας παραγράφου. Η είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Α, τι βλέπω. Λοιπόν, ηλεκτρονική επαλήθευση, γιατί δεν είναι σαφές και ψηφίσω κι εγώ, εκτός εάν δεν επιθυμείτε την ψήφο μου. Οι γυναίκες του ΕΛΚ φαίνονται προβληματισμένες. Τι να συμπεράνω. Τρεις είναι οι δυνατότητες, υπέρ κατά αποχή. Άλλη δεν έχει. Ή μπορείτε να αποχωρήσετε και από την αίθουσα αν θέλετε. Πέρας. Πέρας. 19 υπέρ 16 κατά, καμία αποχή, άρα εγκρίνεται η τροπολογία. Μέσα σε μια γενική σύγχυση, αλλά εγκρίθηκε. 16 στη συνέχεια. Γκέρον και Χάιντερ, εισηγητής κατά, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Ashworth. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Η Γκουε. Άκρος ενδιαφέρον. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18. Των φιλελευθέρων. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Δύο μόνο αποχές εγκρίνεται. Στην παράγραφο 5, τροπολογία 19, Ashworth. Εισηγητής κατά. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Ένας μόνο. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 της Γκουε. Εισηγητής κατά. Υπέρ παρακαλώ. Γκουε και σοσιαλιστές. Κατά. Όλοι οι υπόλοιποι αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 21. Μούλντερ, εισηγητής κατά. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Η ομάδα του Γιάν. Κατά. Πλειοψηφία, αποχές, άρα απορρίπτεται. Στην επόμενη παράγραφο έχουμε την 23 του Ashworth. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Μόνο δύο, α, τρεις έως και τέσσερις. κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 κούε εισηγητής κατά. Υπέρ παρακαλώ. Γκουε και σοσιαλιστές κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 του υποφαινομένου. Ο εισηγητής τίθεται υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Εγκρίνεται. Και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη αυτή. Στη συνέχεια έχουμε τρεις τροπολογίες του Richard Ashworth. Ο εισηγητής είναι κατά. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε από κοινού. Όχι. Όχι. Ωραία. 26. Υπέρ. 2. Κατά. Πλειοψηφία αποχές απορρίπτεται. 27. Υπέρ. 2 μόνο. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23. 28 με συγχωρείτε. Υπέρ. Μόνο 2. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Άσουαρθ και πάλι. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. Ρίτσαρντ Άσχουρθ, επίσης, ο εισηγητής αντιτίθεται. Υπέρ. Ουδής. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31. Μούλτερ. Κατά ο εισηγητής. Υπέρ. Η ομάδα του Γιάν. Συν 2. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32. Richard Ashworth. Κατά ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. 2. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 των σοσιαλιστών. Κατά ο εισηγητής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Οι πράσινοι απέχουν. 34 το υποφαινομένου. Θέλετε να παρουσιάσετε την προφορική, Τζοβάνι. Ναι. Επί της 34 υποβάλλω μια προφορική ζητεί από τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν ώστε οι προβλέψεις που αποστέλουν στην Επιτροπή, με βάση τις οποίες η Επιτροπή προβάλλει τις προτάσεις της για τις πληρωμές, ε, επιβεβαιώνονται σε πολιτικό επίπεδο από όλα τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, επεξήγηση. Επεξηγήσεις. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πολιτικής υφής αίτημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο φτάσαμε με τον εισηγητή στον τριμερή διάλογο εδώ και 15 ημέρες ως προς τις πιστώσεις πληρωμών με τον Υπουργό κύριο Μαύρο Γιάννη και τον Επίτροπο Λεβαντόφσκι από την Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε διαπιστώσαμε ότι η μέθοδος που ισχύει μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για την αποτίμηση των πιστώσεων πληρωμών δεν ήταν η κατάλληλη. Και κάθε χρόνο όταν ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό και μιλάμε για το επίπεδο, επίπεδο πιστώσεων πληρωμών, πάντα Υπάρχουν διχογνωμίες. Η κατάσταση ήταν ε, άκρος δυσάρεστη πέρσι, αν θυμόσαστε. Η έλλειψη σωστής αποτίμησης δημιουργεί ένα θέμα. Κάθε κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο ή σε επίπεδο τοπικό ή εξειδικευμένων οργανισμών που διαχειρίζεται ευρωπαϊκά χρήματα και πιστώσεις για τα προγράμματα συντάσσει τον κατάλογο πιστώσεων πληρωμών που αποστέλει στη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έχει αναλάβει το εν λόγω πρόγραμμα από μέρους της Επιτροπής για το Ταμείο Συνοχής ε, πρόκειται για τη Regio. Για το Lifelong Learning είναι αρμόδια Γενική Επιτροπή Εκπαίδευσης. Η εν λόγω Γενική Διεύθυνση προβαίνει σε τροποποιήσεις, αν το κρίνει σκόπιμο, και το αποστέλει στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμών προβαίνει στις διάφορες τροποποιήσεις, σοβαρές ή μη τροποποιήσεις, κάνει μια αξιολόγηση και προβαίνει στην ε, τελική αποτίμηση. Στις περισσότερες χώρες το Υπουργείο Οικονομικών, τα Υπουργεία Οικονομικών δεν γνωρίζουν ποιες είναι αυτές οι πιστώσεις πληρωμών που ζητούν οι άλλες κυβερνήσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Άρα, εάν ο Επίτροπος ε, Προϋπολογισμών προβάλλει προτάσεις για τις πληρωμές για την επόμενη χρήση, τις υποβάλλει και αν χρειαστεί προβάλλει και διορθωτικό προϋπολογισμό και για την τρέχουσα χρήση. Το σύνολο αυτό που είναι απότοκο αυτών των αλλαγών οδηγεί σε αρνητική αντίδραση των Υπουργείων Οικονομικών που θεωρεί ότι αυτά τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα υψηλά. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρέπει προς τις δαπάνες αυτές, ενώ τα Υπουργεία Οικονομικών ακολουθούν μία άλλη πιο συντηρητική πολιτική. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σκοτεινή πλευρά. Όλα αυτά τα αριθμικά στοιχεία βράζουν σε ένα καζάνι χωρίς να υπάρχει δημοσιότητα προς τα έξω. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος ούτε από τα εθνικά κοινοβούλια, ούτε από το ευρωπαϊκό, που τίθεται ενώπιον τετελεσμένων. Γι' αυτό ακριβώς. Μέσω αυτής της τροποποίησης σας προτείνουμε μία προαπέτηση. Μια διαφορετική, ένα διαφορετικό τρόπο εργασίας και από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη. Να ζητήσουμε από κάθε κράτος μέλος να υπάρχει ένα συγκεντρωτικός χαρακτήρας αποτίμησης των πιστώσεων πληρωμών από όλες τις αρχές που διαχειρίζονται αυτές τις πιστώσεις πληρωμών από πλευράς κράτους μέλους. Ζητάμε μία πιστοποίηση αυτής της διαδικασίας. Για να ξέρουμε ότι αυτές είναι πραγματικές ανάγκες και όχι επίπλαστα στοιχεία τα οποία προβάλλονται για να έχει κανείς περισσότερα κονδύλια. Δημοσιοποίηση αυτών των αριθμητικών στοιχείων στη συνέχεια έτσι ώστε να τα ελέγξουν τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και μετά αποστολή αυτών των αριθμητικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν ισχύσει αυτή η διαδικασία, τι θα κάνει η Επιτροπή, θα προσθέσει τα επιμέρους σύνολα και κανένα Υπουργείο Οικονομικών δεν θα μπορεί να προβάλλει αντιρρήσεις. Διότι ο καθένας θα έχει πιστοποιήσει αυτά τα στοιχεία στην πατρίδα του. Θα υπάρχει δηλαδή μία αρχή ελέγχου και πιστοποίησης η οποία θα ελέγχει αυτά τα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο πρωτίστως. Οι χώρες ε, οι οποίες έχουν ομοσπονδιακό χαρακτήρα ή αποκεντρωμένο δεν το δέχονται αυτό, διότι εκεί η διαχείριση των κονδυλίων, των πιστώσεων αυτών πληρωμών γίνονται από τις τοπικές αρχές. Αυτό ισχύει για την Ισπανία, η Γερμανία και ούτω καθεξής. Και άρα οι τοπικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες. Άρα Πρόκειται για μία διατύπωση που λαμβάνει υπόψη και τις χώρες που έχουν ομοσπονδιακό χαρακτήρα ή πιο αποκεντρωμένο και τις χώρες οι οποίες έχουν ένα συγκεντρωτικό χαρακτήρα διαχείρισης, τρόπο διαχείρισης. Αυτός είναι, αυτό είναι το σκεπτικό που διαπνέει αυτή την προφορική τροπολογία. Με βάση λοιπόν την εισήγηση αυτή, ποιοι είναι υπέρ της τροπολογίας 34. Σας ευχαριστώ. Κατά. Ουδής. Αποχές. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται ομόφωνα λοιπόν η τροπολογία. Τροπολογία υπαριθμών 35 του κυρίου Γκαρίγα. Ο εισηγητή είναι υπέρ, Ποιο είναι υπέρ, κατά. Τρει αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 22 από τους φιλελευθέρους καταπίπτει. Καταπίπτει και η 43 και η 71. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 36 του κυρίου Άσουαρθ. Είναι κατά ο εισηγητής υπέρ. 2 κατά. Οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 37 της ΓΚΟΕ. Κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλγα. Απορρίπτεται. Τροπολογία 38. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Φιλελεύθερη. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Εδώ έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα, τρία τμήματα, μας το έχουν στήσει φιλελεύθεροι. Αυτό πρώτο τμήμα ξεκινάει με το Underlines Done έως Rebuild Confidence in the Economy. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. Τρεις. Αποχές. Καμία εποχή εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ξεκινάει με το «Has already been critical» έως «Reduce them down to 1.27 compared to budget» υπέρ. Κατά. Φιλελεύθερη και η FD αποχές. Μία αποχή εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. EFD, αποχές, εγκρίνεται. Εγκρίνεται λοιπόν το σύνολο της συμβαστικής τροπολογίας, πράγμα που σημαίνει ότι καταπίπτουν οι επόμενες τροπολογίες έως την προφορική τεχνική τροπολογία του Τζοβάνι Λαβία. Είναι καθαρά τεχνική η τροπολογία αυτή, δεν προβλέπεται ψηφοφορία, προς ενημέρωσή σας απλώς περιλαμβάνεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 44 του κυρίου Άσχορθ κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 45 της Γκουε κατά ο εισηγητής υπέρ. Μόνο η Γκουε κατά. Οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 46. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες κατά ο εισηγητής υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την τροπολογία 46. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πρέπει να είστε υπέρ, αλλά θα το επαληθεύσουμε. Έχετε όλοι τις κάρτες σας, ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 18 κατά μία αποχή, επομένως απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 47, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ, κατά. Τρεις αποχές εγκρίνεται. Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 48 καταπίπτει, όχι όμως και το δεύτερο. Επομένως ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 48 κατά ο εισηγητής υπέρ. Ουδής, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 49, της ο εισηγητής είναι υπέρ, εφόσον προσθέσουμε end jobs και θέσεις εργασίας. Είναι υπέρ της δημιουργίας θέσεων εργασίας η Γκούε υπέρ, κατά, ένας, αποχές, εγκρίνεται. Στη συνέχεια έχουμε μία τεχνική τροπολογία στην παράγραφο 19 του Τζοβάνι Λαβία. Δεν προβλέπεται ψηφοφορία για αυτήν. Περνάμε λοιπόν στις τροπολογίες 50 και 51 της Έλγα Τρούπελ που θα τις ψηφίσουμε από κοινού. Υπέρ παρακαλώ. 4. Κατά. Οι περισσότεροι αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 52 της Έλγα Τρούπελ κατά η εισηγήτρια υπέρ. 4 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 της Μπάρμπαρα Ματέρα υπέρ εισηγήτρια, υπέρ, κατά, αποχές, φιλελεύθερη και πράσινη και ο κύριος Άτογκ, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 54 την έχει αποσύρει η Μπάρμπαρα. Μάλιστα. Τροπολογία 55, Σαλβαδόρ Γκαρίγα. Υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Οι σοσιαλιστές και η Έλκα αποχές. Σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 56. Ντομινίκ Ρικέ με προφορική τροπολογία του εισηγητή προκειμένου να διαγραφεί η φράση calls for maintaining και να πούμε therefore decides to maintain. Συνεπώς αποφασίζει να διατηρήσει. Είναι πιο στεναρό αυτό. Υπέρ. Κατά. Ένας. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη παράγραφος, τροπολογία 57 του Ρίτσαρτ, κατά ο εισηγητής, υπέρ. 2. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 58 της Γκουε. Μας κάνει εντύπωση, ότι είναι υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Η φιλελεύθερη, η ευτή, άρτονγκ, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 59, που είναι συμβατή, του Γιάν Μούλντερ, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ, κατά. Τρεις, αποχές, εγκρίνεται. Επόμενη παράγραφος, νέα, τροπολογία 60 του κύριου Φερέιρα, κατά ο εισηγητής υπέρ. Δύο, Κατά. Οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 61 του Ρίτσαρτ, ο εισηγητής είναι κατά, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Επόμενη παράγραφος. Τροπολογία 62 του Ρίτσαρντ Άσχορτ ε, κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 63 της Γκουε υπέρ ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Φιλελεύθερη FD Αρτόγκ. Αποχές εγκρίνεται. Φτάσαμε στη βαστική τροπολογία παριθμών 3 για την παράγραφο 24. Υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Άρα μπορούμε να περάσουμε αμέσω στην τροπολογία 67 του Ρίτσαρτ Άσχορθ κατά ο εισηγητής υπέρ. Τρεις κατά, οι περισσότεροι, αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη, απορρίπτεται λέει ο Πρόεδρος. Τροπολογία 68, υπέρ ο εισηγητής, υπέρ κατά, δύο αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 69. Ρίτσαρτ Ashworth. Ο εισηγητής είναι κατά υπέρ. 3. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 70 του ίδιου εισηγητή κατά ο εισηγητής υπέρ. 4 κατά. Οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 27. Έχουμε πάλι μια προφορική τροπολογία τεχνικής φύσεως του Τζοβάνι, δεν την ψηφίζουμε. Περνάμε στην 72 της Έλκα Τρούπελ, κατά εισηγήτρια υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επόμενη παράγραφος, τροπολογία 73 του Ρίτσαρτ, κατά ουσηγητής υπέρ. 3. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74. Διντεργεράν υπέρ ο εισηγητής ποιος είναι υπέρ, κατά, η φιλελεύθερη, η ευτή και ο κύριος Άρτογκ, αποχές εγκρίνεται. Επόμενη παράγραφος, τροπολογία 75 του κυρίου Φερέιρα, κατά ο εισηγητής υπέρ. 3. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 76. Εδώ έχουμε χωριστή ψηφοφορία κατά τμήματα που έχουν ζητήσει οι εισηγητές της τροπολογίας. Στο πρώτο τμήμα επιθυμούν μία διαγραφή, μάλλον διαγραφή του πρώτου τμήματος. Realistic approach. Υπέρ αυτού του πρώτου τμήματος. Κατά αποχές επομένως απορρίπτεται. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο τμήμα, δηλαδή μάλλον τη διαγραφή του δεύτερου τμήματος, τις τροπολογίες από το Considerous μέχρι το Agricultural Policy, υπέρ ο εισηγητής, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, άρα το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας εγκρίνεται, μάλλον θα διαγραφεί ουσιαστικά. 77 της κυρίας Τρούπελ κατά εισηγήτρια υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 της Γκούε κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ, νομίζω ότι περισσότεροι είστε κατά, αλλά σε επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για την τροπολογία 78, άρτη ψηφοφορία, κατά ο εισηγητής. Πέρας. 14 υπέρ, 22 κατά, καμία αποχή. Όντως λοιπόν απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 79 του Ρίτσαρτ Άσχουαρθ Κατά είναι ο εισηγητής, ποιος είναι υπέρ. 2. Κατά. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Ναι, κατά. Αποχές. Οι περισσότεροι είναι κατά λοιπόν. 80 του Ρίτσαρτ Άσχορθ, ο εισηγητής είναι κατά, υπέρ. Τρεις, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 81. Γκαρτέν και Γκεράν, υπέρ, εισηγητές, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 του Ρίτσαρτ Άσχορθ, κατά, ο εισηγητής, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 83 της Έλγα Τρούπελ, η εισηγήτρια είναι κατά, υπέρ. Τρεις, νομίζω, να σας μετρήσω. Εννέα, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 84 των φιλελευθέρων. Υπέρ ο εισηγητής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τέσσερις αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 85 του κύριου Γκέρμπραντι Υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Τρεις αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 86 η οποία είναι συμβατή. Είναι κατά ο υπέρ. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στις πολιτικές ομάδες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14 υπέρ, 22 κατά. Καμία αποχή απορρίπτεται λοιπόν. Γυρίζουμε σελίδα, περνάμε στροπολογία 87. Μπορούμε τις 87 και 88 να τις ψηφίσουμε από κοινού. Είναι κατά ο εισηγητής. On block ψηφίζουμε πάντως, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Επόμενη παράγραφος, Στροπολογία 89 του Ρίτσαρτ. Ο εισηγητής είναι κατά, υπέρ. Δύο κατά. Οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται. Στην ίδια παράγραφα έχουμε τροπολογία 90 της ΓΚΟΕ κατά ο εισηγητής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 91 της Έλγα Τρούπελ κατά εισηγήτρια υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η ίδια με την προηγούμενη τροπολογία. Τροπολογία 92 του Ρίτσαρτ Άσχορθ κατά ο υπέρ. 3. Κατά. Οι περισσότεροι. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 93 της Γκουε κατά ο εισηγητής υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 94 του Αλεξάνδρα Άλβαρο κατά είναι ο υπέρ. η ομάδα του κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία παριθμών 4 για την παράγραφο 40 υπέρ της συμβαστικής τροπολογίας κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη τροπολογία 99 έιντερ κατά ο εισηγητής υπέρ. Η πολιτική του ομάδα και η Γκουε κατά οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 100 του Ρίτσαρτ Άσχορθ κατά ο συγητής υπέρ. 3. Κατά. Οι περισσότεροι αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 101 του Ρίτσαρτ κατά ο συγητής υπέρ. 2. Κατά. Αποχές. 1, Αποχή και απορρίπτεται. Τροπολογία 102 της Μπάρβαρα Ματέρα, η εισηγήτρια υπέρ, υπέρ. Κατά. 3. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν, μάλλον η 103 είναι συμβατή ή όχι. Είναι συμβατή. η τροπολογια Σέιντερ και Ματέρα, Μπάρπαρα Ματέρα είναι συμβατές. Ψηφίζουν 103 υπέρ, κατά. Δύο αποχές. Εγκρίνεται η 103. Γυρίζουμε σελίδα. Τροπολογία 104 του Ρίτσαρτ Τάσχορθ κατά ο συγητής υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 105 έχει αποσυρθεί. Έτσι δεν είναι. Πάμε στην 106 την οποία έχουμε διατηρήσει. Μπορούμε να ψηφίσουμε από κοινού την 106 και την 107. Όχι. Λοιπόν, την 106 υπέρ ο εισηγητή, υπέρ. Κατά. Η φιλελεύθερη, η FD και ο κύριος Σάρτονγκ. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 107 υπέρ. Κατά. η ίδιοι συν την ΕΛΓΑ, οι περισσότεροι είναι υπέρ, αποχές εγκρίνεται. Φτάνουμε στη βασική τροπολογία υπαριθμών 5 υπέρ, κατά, τρεις αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 111, έντερ, υπέρ ο συγητής, υπέρ, κατά. Δύο αποχές, εγκρίνεται. 112 του Ρίτσαρτ Άσχορθ, κατά ο συγητής, υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 113 της Γκουε, κατά ο εισηγητής υπέρ. 2 κατά πολύ αποχές και απορρίπτεται. 114 του Ρίζα Τάσχορθ κατά ο εισηγητής υπέρ. 1 κατά αποχές απορρίπτεται. 115 Έιντερ υπέρ ο εισηγητής υπέρ κατά ένας αποχές εγκρίνεται. Επόμενη παράγραφος. Εδώ έχουμε μία τροπολογία προφορική τεχνικής φύσης που δεν θα την ψηφίσουμε όμως. Θα ψηφίσουμε όμως την 116 του Richard Ashworth. Μπορούμε την 116, 117 και 118 να ψηφίσουμε μαζί. Όχι μου λένε. Μόνο την πρώτη λοιπόν. 116 κατά ο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 117 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ. Ένας κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μπορούμε την 119, 120, 121 ψηφίσουμε από κοινού. Πολύ ωραία. Υπέρ. Κατά ο εισηγητής. Όχι, δεν θέλετε από εκείνο να ψηφίσουμε. Μάλιστα, λοιπόν, 119 υπέρ. Ένας κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. 7. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έχει αποσυρθεί η τροπολογία 122. Σωστά πληροφορούμε. Ναι. Είχαμε συμπεριλάβει την τροπολογία αυτή στην προηγούμενο ψήφισμα. Θα, θα προτιμούσα πάντως να την ψηφίσουμε, γιατί δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Γκερμπράντι ακόμα. Ας την ψηφίσουμε λοιπόν, αν γίνει τώρα. Την ψηφίσουμε υπέρ ο εισηγητής. Υπέρ. Κατά. Σοσιαλιστέ και Δημοκράτες αποχέ και ο κύριο Σέρκτονγκ Αποχέ εγκρίνεται. Ενδιαφέρουσα περίπτωση μια τροπολογία που έχει αποσυρθεί αλλά παρόλα αυτά είναι κρίθη. 123. Τρίπελ. Ο συγκητής κατά. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Τρει κατά. Η πλειονότητα απορρίπτεται. 124 των φιλελευθέρων. Ο συγκητής είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 125. Χάουγκ. Με προφορική τροπολόγηση του εισηγητή. Ο εισηγητής. Η προφορική αφορά την εισαγωγή ορισμένων παραδειγμάτων αποκλειστικά. Is ότι γνωρίζει ότι ορισμένοι οργανισμοί, εγώ θα ήθελα να ε, αναφερθούμε στη Europol, να κλείσουμε την παρένθεση και την ΑΖΕ ΑΣΕΡ. Δηλαδή να βάλουμε ορισμένα παραδείγματα αναφερόμενοι στους οργανισμούς και να κλείσει η παρένθεση. Ωραία. Συμφωνεί ο υποβάλλον την τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας με την προφορική συμπλήρωση, κατά, αποχές εγκρίνεται 126 Ashworth ο συγκεκριτής είναι κατά υπέρ 3 κατά αποχές απορρίπτεται να περάσουμε τώρα στο τμήμα που αφορά τα άλλα θεσμικά όργανα Άρα τον άλλο εισηγητή. 127. Γκέραν. Εισηγητής είναι υπέρ. Ποιοι άλλοι είναι υπέρ. Κατά. Τρεις. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 φιλελευθέρων. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται επίση. 129 το ΕΛΚ έχει ζητήσει ε, ψηφοφορία κατά τρία τμήματα. Είναι η τροπολογία στην οποία αναφέρθηκε ο Ντέρεκ προηγουμένως. Αν θα έρθει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Στρασβούργο ή όχι. Ο εισηγητής προτείνει ε, ε, ελευθερία ψήφου. Για το πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά να ελέγξουμε. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. 16 υπέρ, 18 κατά, απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Πέρας. 19 εννέα υπέρ, δεκατέσσερις κατά μία αποχή, εγκρίνεται το τρίτο τμήμα. Ωραία. Να περάσουμε τώρα στην επόμενη συμβαστική. Συμβαστική 6, μείον την 136. Ωραία. Κέραν. Μπορεί να απογοητεύσει τον κύριο Χάτον, αλλά όπως είπα και στον εισηγητή είμαι υπέρ της συμβαστικής. Άρα εάν εγκρίνουμε τη συμβαστική θα αποσύρω την 136. Ωραία λέει ο πρόεδρος. Αλλά κύριε Χάρτον, κύριε Χάρτον, αν αποσυρθεί από τον συντάκτη της η τροπολογία, έχετε δυνατότητα να την επανυποβάλλετε. Εάν επιθυμείτε. Ωραία. Θα ψηφίσουμε χωριστά λοιπόν αυτή την τροπολογία. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 6 εκτός της τροπολογίας 136. Ποιοι είναι υπέρ της συμβαστικής 6. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 136 τώρα που δεν είναι πλέον του Γιώργου αλλά του κυρίου Χάρτον. Ποιοι είναι υπέρ. Τροπολογία 136. Είστε υπέρ βεβαίω. Και ε, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία. Οπότε περνάμε τώρα την 135 του Ντέρεκ επί της οποίας έχει μια προφορική τροπολόγηση ο Ντέρεκ. Α, που είναι στο κείμενο. Έχετε το κείμενο μπροστά σας. Είναι τεχνική. Αλλάζουμε το, το πάγωμα σε ε, τη μαθηματική αναψαρμογή. Ποιοι είναι υπέρ. Είναι τεχνική τροπολογία. Κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε, τώρα περνάμε στην παράγραφο 83 Υπάρχει η προφορική τροπολογία του κυρίου Φέρμ να αντικαταστήσουμε τη λέξη αεροπορικές εταιρείες με αεροπορικά εισιτήρια. Θα την κάλυπτε η 136, αλλά απορρίφθηκε. Άρα πρέπει, άρα πρέπει να ψηφιστεί. Ο συγητής είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 137. Lion. Έχει αποσυρθεί. Α, ωραία. 138 και 139 του Γκέραν μαζί. Όχι, όχι. Καλά. 138. Ο συγητής είναι υπέρ. Υπέρ ποια άλλη είναι. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη. 14 υπέρ, 20 κατά. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 139, ο συγκητής υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά η φιλελεύθερη, ο κύριος Χάρτον, αποχές, η Έλγα, απέχει, εγκρίνεται. Τρεις τροπολογίες Ashworth, μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Πολύ ωραία. Ο συγητής είναι κατά. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Τρεις. Κατά η πλειοψηφία. Αποχές απορρίπτονται. 143 έλγα. Ο συγητής είναι κατά. Υπέρ. Τρεις. Κατά η πλειοψηφία. Αποχές απορρίπτεται. Οι τρεις τελευταίες τροπολογίες. Άσουετ, μπορούμε να τι ψηφίσουμε μαζί. και είναι υπέρ. Τρεις. Κατά. Η πλειοψηφία. Αποχές. Απορρίπτονται. Οπότε. Ως παράρτημα θα επισυνάψουμε τις γνωμοδοτήσεις όλων των επιτροπών που κλήθησαν να γνωμοδοτήσουν και θεωρούμε ότι όλες αυτές οι γνωμοδοτήσεις καλύπτονται από τις ψηφοφορίες που κάναμε εδώ στην Επιτροπή μας ή καταπίπτουν λόγω των ψηφοφοριών μας. Και το σύνολο θα επισυναυθεί στο ψήφισμά μας, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του ψηφίσματος. Άρχεται. Ψηφίστε παρακαλώ. Ωραία. Πέρας. 27 υπέρ, 2 κατά 5 αποχές. Συγχαίρουμε τους δύο εισηγητές μας για την ε, θαυμάσια εργασία τους, που είναι η επιβράβευση μηνών εργασίας και η κατάληξη των ψηφοφοριών επί των ε, στοιχείων και των σχολείων και των τροπολογιών της προηγούμενης εβδομάδας. Θα συνεχίσουμε να ψηφίζουμε. Α, όχι. Οι άλλες ψηφοφορίες θα γίνουν το απόγευμα. Διότι για το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση δεν είναι έτοιμες όλες οι πολιτικές ομάδες. Πέρας των ψηφοφοριών για σήμερα το πρωί λοιπόν και να περάσουμε στην ε, συζήτηση, την συνέχιση της συζήτησης για την ενδιάμεση έκθεση. Οι κύριοι εισηγητές, ο Ράινα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήδη τη Δευτέρα το απόγευμα μεταξύ ο λιγότερων κάναμε μια πρώτη συζήτηση για αυτή την ενδιάμεση έκθεση Έχουν υποβληθεί 202 τροπολογίες και μετά τη συζήτηση τη Δευτέρα ο Ήβαλο και εγώ προσπαθήσαμε να καταλήξουμε στους αναγκαίους συμβιβασμούς όπως και για τους ίδιους πόρους η Ντεάν και Γένσεν γιατί είναι τμήμα της έκθεσής μας ε, αυτά που συζήτησαν εκείνοι τη Δευτέρα το απόγευμα λοιπόν και την Τρίτη είχαμε δύο συζητήσεις με στόχο όσο ήταν δυνατόν να συμπεριλάβουμε τις ε, τροπολογίες χωρίς να θίξουμε τους βασικούς προσανατολισμούς της έκθεσης. Έχουμε λοιπόν 27 συμβαστικές ε, τροπολογίες που τις έχετε και μερικές προφορικές. Να επαναλάβω σαφώς το εξής. Αυτή η ενδιάμεση έκθεση με βάση τον κανονισμό μας έχει στόχο η διαδικασία έγκριση των ε, πολιετών δημοσιονομικών προπτικών να επιταχυνθεί, να διευκολυνθεί και μετά από την ψηφοφορία ε, στις 20 Οκτωβρίου στην ε, Επιτροπή και στην Ολομέλεια θα προσφερθεί στην Προεδρία του Συμβουλίου ούτω ώστε να καταλάβουν ότι είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε μια συμφωνία για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο επειδή βεβαίως η διαδικασία και από πλευρά του Συμβουλίου έχει επιταχυνθεί. Βέβαια δεν ξέρουμε που θα καταλήξει, αλλά επειδή θα υπάρξει στις 22 και 23 Νοεμβρίου το ειδικό Συμβούλιο Κορυφής, πρέπει η έκθεσή μας να βοηθήσει τη διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τα κεντρικά σημεία που μαζί εκπονήσαμε με βάση τις προηγούμενες εκθέσεις το θέμα της συμπερίληψης της στρατηγικής 2020 για ανάπτυξη και απασχόληση, την τάξη μεγέθους που θέλουμε για, τα, για τις δαπάνες, το θέμα της καλύτερης ε, δαπάνησης, το θέμα κατά πόσο πρέπει να δίνουμε σε άλλους φορείς τα μεγάλα προγράμματα, τη διάρκεια δηλαδή πότε θα χρειαστεί να γίνει η αναθεώρηση στη μέση της περίοδου, να έχουμε ένα καλύτερο λοιπόν δημοσιονομικό πλαίσιο, μιλήσαμε και για την ενότητα του προπολογισμού και κυρίως για τους ιδίους πόρους. Αυτό βεβαίως δεν αποκλείει, ανάλογα με το πώς θα αντιμετωπιστεί η προσφορά μας αυτή, από προεδρίας, από πλευράς προεδρίας, και ανάλογα με το πώς θα προχωρήσει και ο κύριος Φανρόμποη. Μπορεί λοιπόν να υποβάλουμε συμπληρωματικό ψήφισμα, να χρειαστεί ενδεχομένως να υποβάλουμε συμπληρωματικό ψήφισμα για την έκτακτη συνάντηση κορυφής του Νοεμβρίου, ούτω ώστε να καταστήσουμε σαφή τα όρια μας, τις κόκκινες γραμμές μας, αλλά είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε, θέλουμε να καταλήξουμε σύντομα, αλλά δεν θα πρέπει λόγω της ταχύτητας διαπραγμάτευσης να θυγεί η ποιότητα των προσπαθειών μας, αλλά είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο μέχρι το τέλος του χρόνου. Παράλληλα όμω, πρέπει και από πλευρά του κάτι να κάνουν. Οι τροπολογίε μα, οι συμβαστικές, έχουμε, έχουν στόχο να επιτύχουν όλους αυτούς τους στόχους. Κατάλληλη χρηματοδότηση, ποιότητα της δαπάνησης ε, Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει παραλληλισμός μεταξύ του πλαισίου και των πολιετών προγραμμάτων. Θέλουμε ευληγησία του χρόνου εφαρμογής, γιατί όσο πιο περίπλοκα είναι τα ε, ε, αριθμητικά στοιχεία, τόσο περισσότερη ευληγησία χρειάζεται στον τρόπο δαπάνησης τους. Και επίσης θέλουμε να υπάρξει ε, ξεμπλοκάρισμα και της κατάστασης στους ιδίους πόρους. Ε, δεν ξέρω αν και ο συνάδελφος ε, Κάλφιν θέλει το λόγο, αλλά θα ήθελα ακόμη να πω ότι υπήρξε θαυμάσια συνεργασία και η βοήθεια της γραμματείας και οι σύμβουλοι επίσης μας βοήθησαν πάρα πολύ. Αλλά επειδή ο κόσμος ε, δεν συνεχίζει να κινείται, μπορεί να μας εκπλήξουν περαιτέρω εξελίξεις, αλλά πρέπει να μείνουμε στους στρατηγικούς μας προσανατολισμούς. Είδατε ότι η ομάδα εργασίας των Προέδρων μιλάει για προϋπολογισμό για την Ευρωζώνη. Και παρατηρούμε επίσης τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου να το εγκρίνει αυτό για προφανείς λόγους, αλλά υπάρχουν κράτη-μέλη που επιδιώκουν αυτήν την διέξοδο όταν ε, είδαν τι έγινε με την εφαρμογή του ΒΕΤΟ, όταν προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε τη φορολογική διάσταση στην Ευρωπαϊκή ε, Συνθήκη, για να μην υπάρχει μονίμως αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτή η πρακτική δημιουργεί και πολλά προβλήματα. Διότι η σκέψη ότι εκτός από την κατοχήρωση και τη δημοσιονομική πειθαρχία να κάνουμε και κάτι άλλο για την Ευρωζώνη, είναι βέβαια συναρπαστική πρόκληση. Δεν πρέπει να αποκλείουμε αυτή την προσπάθεια. Υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο και κυρίως ο Πρόεδρος μας επέμεναν ότι τα 60 δισεκατομμύρια που ήταν στον πρώτο προπολογισμό για τη διάσωση έπρεπε να μπουν με ένα προς υπόμνηση. Έχουμε δηλαδή στον προπολογισμό μας στοιχεία για τον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Γιατί λοιπόν να μην το επεκτείνουμε αυτό, τίθεται το ερώτημα. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, γιατί υπάρχουν πολλέ παράλληλε δραστηριότητε σε, αυτό, σε αυτή την ομάδα εργασία όπου έχει προσκληθεί ως, ε, ε, ως προσκεκλημένος και ο πρόεδρος Σούλτς. Παράλληλα όμως συνεχίζουμε τις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Διότι δεν είναι δυνατόν να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα όταν μειώνουμε τα ποσά στο πολιετές πλαίσιο και όταν ε, μας λένε επίσης ότι ανάλογα με το πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις για το πολιετές πλαίσιο μπορεί να κάνουμε και κάποιες συζητήσεις για τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Δεν είμαι νομομαθής, αλλά πιστεύω ότι κάτι τέτοιο παραβιάζει βασικές αρχές των ευρωπαϊκών συνθήκων. Το ευρώ είναι η συνήθις περίπτωση των ε, συνθήκων. Και η μη συμμετοχή στην Ευρωζώνη είναι η εξαίρεση. Και όλες οι χώρες που το επιθυμούν και που δεν αξιοποιήσουν αυτή την εξαίρεση, ευχαρίστως εάν ε, πληρούν τις συνθήκες, να εισέλθουν στη ζώνη ευρώ. Αυτή η συζήτηση που γίνεται στη συζήτηση και που δεν μπορώ να αποτιμήσω που θα καταλήξει, πρέπει να μας καλέσει να καταλάβουμε τι επιπτώσεις έχει η στρατηγική και οι θέσεις μας. Δεν είναι δυνατόν η συνήθις περίπτωση, δηλαδή ένα ισχυρό ευρώ στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς όπου συμμετέχουν 17 χώρες και άλλες θα μπουν όταν ε, πληρούν τις συνθήκες, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να θεωρηθούν ως ε, παράπλευρο στοιχείο και να θεωρηθεί ότι το πιο ασθενές κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κύριο. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν προωθεί την ευρωπαϊκή ενοποίηση και θα ήταν η αρχή περαιτέρω διακυβερνητικοποίησης. Οπότε θα τεθούν θέματα και δημοκρατικότητας της διαδικασίας και τήρησης των αρχών της Λισαβόνας, της συνθήκης της Λισαβόνας. Γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα εκφραστούμε Ίσως όχι μέσω ενός ε, επιπλέον ε, ε, μέσω μιας επιπλέον τροπολογίας, αλλά πιστεύω ότι οι ομάδες θα έπρεπε να σκεφτούν πώς μπορούν να διευκρινίσουν ότι είναι υπέρ και της ενότητας του προπολογισμού μέσω της τροπολογίας 175, αλλά ενδεχομένως να το συμπληρώσουμε και με κάποια κείμενα στα παραρτήματα και όλα αυτά διότι εάν δεν ε, αναλάβουμε αυτές τις ενέργειες θα έχουμε μετά μεγάλες δυσχέρειες για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις αυτής της νέας δυναμικής που μοιάζει να διαφαίνεται. Μετά την ψηφοφορία θα ήθελα θα ήθελα να θέσω στο παράρτημα ένα κείμενο της ομάδας εργασίας μου για τις πολιετής προοπτικές για να καταστεί σαφές ότι ήδη από σήμερα είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε σε οτιδήποτε προκύψει και να προωθήσουμε ταχαίως τις διαπραγματεύσεις με την Προεδρία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σίγητα. Ο Ήβαλο. Ευχαριστώ πρόεδρε ορισμένα επιπρόσθετα σημεία. Καταρχήν να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και τους πολιτικούς ε, συνομιλητές και συμβούλους, διότι μας βοήθησαν να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και όλες τις άλλες πολιτικές ομάδες, τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες. Στις, στους συμβιβασμούς αυτούς βλέπετε ότι επήλθαν πολύ δύσκολες συμφωνίες μετά από μια κατάσταση δυστοκίας θα μπορούσα να πω. Προσπαθούμε να φτάσουμε στην ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Αυτό είναι κάτι ύψης της σημασίας από πλευράς του Κοινοβουλίου. Επίσης, αρκεστήκαμε στα δεδομένα της Επιτροπής ε, ΣΥΡ και στο γεγονός ότι τα κείμενα αυτά θα πρέπει να σχετίζονται με το ίδιο το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν θέματα συναπόφαση, τα περισσότερα δηλαδή, προσπαθούμε όμως να τα ελαχιστοποιήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τις δικές σας αντιδράσεις. Νομίζω ότι τα περισσότερα θέματα που είχαν θυγεί περιλαμβάνονται στο συμβιβασμό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες που υπέβαλαν ε, συμβιβασμούς γιατί ε, βελτιώνουν την έκθεση. Σε σχέση με αυτά που είπε ο Ράιμερ, εργαζόμαστε για το επόμενο MFF μετά ή κατά τη διάρκεια φημών ότι προετοιμάζεται ένας νέος κοινοτικό προπολογισμό. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Εάν θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, δηλαδή ότι 11 χώρες έχουν ζητήσει επιταχυμένη διαδικασία για την έγκριση του προϋπολογισμού και, τον ε, και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις προσόδους. Εάν θα ενταχθούν σε αυτόν τον προϋπολογισμό που συζητούμε ή όχι, ή σε άλλους. Όλα αυτά σχετίζονται με το MFF. Όλες αυτές οι ιδέες βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που ήδη εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση και είναι μία πρωτοβουλία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι σε αυτή την έκθεση και σε άλλες που θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα, με βάση την έκθεση Τίσεν, θα πρέπει να αρκεστούμε στην κοινοτική μέθοδο και να εμείνουμε σε αυτήν γιατί διαφορετικά το MFF θα βρίσκεται στον αέρα, αν δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μία δίστοκη συνεργασία. Ευχαριστούμε Ήβαλο. Ζαν Λουίκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι εργαστήκαμε σε θέματα συνολικών πόρων. Έχουμε υποβάλει αρκετές προτάσεις και όπως θα γνωρίζετε, πρόθεσή μας σε αυτή την έκθεση ήταν να ορίσουμε καλύτερα πώς μπορούμε να προσδώσουμε περισσότερα επιχειρήματα στο MFF, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο εξού και τα 5-6 σημεία στο ψήφισμα. Θα ήθελα όμως να συμφωνήσω με τους δύο εισηγητές, γιατί όταν μιλάμε για τους τελικούς πόρους, αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, καθέφτο, γιατί 11 χώρες προσυπέγραψαν αυτή τη συνεργασία, τη συνεργασία επιταχυμένης συνεργασίας, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα προωθηθεί αυτή η συνεργασία. γιατί πολλοί θέλουν να χρησιμοποιήσουν την επιταχυμένη διαδικασία συνεργασίας για να ε, χρηματοδοτήσουν τους επιμέρους προϋπολογισμούς. Άρα αυτό υποσκελίζει τις τελικές προτάσεις ως προς το MFF, το πολιετές δημοσιονομικό. Θα πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν, γιατί μιλάμε για προϋπολογισμούς της Ευρωζώνης και θα μπορούσαν αυτοί οι προϋπολογισμοί να επηρεάσουν την ε, συνολική συζήτηση. Επίσης, μίλησα για τις προτάσεις μας τις έχω εντάξει σε ένα έγγραφο, ως προς τους ίδιους πόρους από το ΦΠΑ. Θέλουμε να τονίσουμε την επιθυμία μας ώστε ένα μέρος του ΦΠΑ να παραμείνει στους ίδιους πόρους. Αν και υπάρχει μια τάση στο Συμβούλιο περί διαγραφής. Γι' αυτό προβάλλουμε και αυτή τη γνώμη ως προς το ε, ΦΠΑ που θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ιδίων πόρων. Επίσης ε, θεωρώ ότι και η Ράιμερ και, ότι η Ράιμερ και Ήβαλο είχαν ένα πολύ δύσβατο και δύσκολο έργο και εν πάση περιπτώσει δεν θα ε, επαναλάβουμε τα λεγόμενα της Επιτροπής ΣΥΡ στην έκθεση αυτό. Ως προς τους ίδιους πόρους ε, δεν θα ήθελα να προσθέσω πολλά σε σχέση με αυτά που είπε ο Ζαν Λουκ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ε, πολιτική μας, την πολιτική συμφωνία που ζητήσαμε. Είπαμε ότι δεν θα συνενέσουμε στο πολιετές δημοσιονομικό εάν δεν συμφωνήσουμε ως προς τις, τους ίδιους πόρους. Αυτό αναφέρεται στο 59 με τα 6 σημεία και και εάν δεν φτάσουμε σε αύξηση των ιδίων συγγνώμη, μείωση των ιδίων πόρων με βάση το ΑΕΠ, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να προβάλλει επιπρόσθετες προτάσεις για τους ίδιους πόρους. Και ζητούμε να φτάσουμε στην μείωση των εθνικών συνεισφορών ως προς την, τους ίδιους πόρους. Ε, η σύνταξη είναι ιδιαίτερα ευτυχής και θα ήθελα την υποστήριξη όλων. Ευχαριστούμε και ευχαριστούμε και στους δύο εισηγητές. Σαλβαδόρ Γκαρίγα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φαντάζομαι ότι μερικοί συνάδελφοι θα έχουν ε, ιδιαίτερα προβλήματα με αυτές τις τροπολογίες συμβιβασμού. Θα ήθελα να πω ως πολιτική ομάδα, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τους τεσσάρους συναδέλφους που συνέταξαν τις εκθέσεις αυτές. Αποτελεί μια στεναρή διαπραγματευτική βάση για τις διαπραγματεύσεις μας με το Συμβούλιο Ακολουθούμε τη γραμμή ΣΥΡ, της Επιτροπής ΣΥΡ, όπως ε, ορίστηκε το 11, ενημερώνει τα στοιχεία, τα επικαιροποιεί και επιτρέπει μια ρεαλιστική διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Δηλαδή μιλάμε για μείωση των αρχικών αριθμητικών στοιχείων της πρότασης Επιτροπής και νομίζω ότι βρίσκουμε εναλλακτικές όδους άσκησης πίεσης προς το Συμβούλιο, ιδιαίτερα ως προς την, τις χρηματοδοτήσεις εγγραφής των και ευελιξία, γιατί δεν έχουμε αρκετούς πόρους για την εκτέλεση των κοινοτικών προγραμμάτων και γι' αυτό θα πρέπει ο προϋπολογισμός να είναι κατά το δυνατόν ευέλικτος. Άρα η ευελιξία είναι ένα πολιτικό ζήτημα, αλλά έχει και την τεχνική της υφή. Γι' αυτό συμφωνώ με τα δεδομένα της έκθεσης. Θα ήθελα να ζητήσω από τις άλλες πολιτικές ε, ομάδες να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με βάση αυτούς τους συμβιβασμούς αποτελούν μια κοινή απαρχή. Πολλοί μπορεί να μην συμφωνούμε με αυτές τις παραγράφους, αλλά εν πάση περιπτώσει η έκθεση αυτή θα πρέπει να ακολουθήσει αυτή τη διάρθρωση δηλαδή των συμβιβασμών και να μην φτάσουμε, προχωρήσουμε σε μεμονωμένες τροπολογίες που δεν θα μπορέσουν να υποστηρίξουν οι άλλες πολιτικές ομάδες και θα μπορούσαν να αποπροσανατολίσουν αυτή την συνενετική διαδικασία την οποία χτίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ, η κυρία Τρούπελ. Σε ευχαριστώ, αλλά. Καταρχάς, να καταστήσω σαφές ότι κοινό μας στόχος πρέπει να είναι να υπάρξουν περισσότερα, περισσότεροι ήδη πόροι για την Ένωση για να γίνει πιο ανεξάρτητη. Αυτό νομίζω ότι μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Να καταστήσουμε επίσης σαφές, τώρα που θα αρχίσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις, ότι ως Κοινοβούλιο, αλλά και η κοινή γνώμη πρέπει να το καταλάβει αυτό, να καταστήσουμε λοιπόν σαφές ότι δεν πρόκειται να παίξουμε το παιχνίδι, όπου οι διαπραγματεύσει για το πολιετέ πλαίσιο, όπου έχουμε βεβαίω κάποιο δίκαιο και δεν πρέπει να το καταλήψουμε, να περιοριστούν διότι μπορεί να συνδυαστεί με, με μια συζήτηση για χωριστό προϋπολογισμό της ε, Ευρωζώνης. Αυτό οπωσδήποτε θα γίνει με νέα διακυβερνητική ε, διάσκεψη όπου θα είναι περιορισμένη η δυνατότητα παρέμβασης και θα μειωθούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Ενώ λοιπόν όλοι θέλουμε να υπάρχει περισσότερη δημοκρατία, ότι πρέπει εμείς πρέπει να ελέγχουμε περισσότερο τον προπολογισμό, υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί μια περιοχή όπου δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα παρέμβασης. Διάβασα τα εξή στον ε, ε, Ευρωπαρατηρητή σήμερα. Το σχέδιο για τη συνάντηση κορυφή, το σχέδιο τη ε, ημερήσια διάταξη προτείνει ένα χωριστό προπολογισμό για την Ευρωζώνη. Τα τελευταία πορίσματα ε, ενώπιον τη ε, συνάντηση κορυφή επόμενη εβδομάδα διαχωρίζουν τον προπολογισμό τη Ένωση από τον προπολογισμό τη Ευρωζώνη. Και ένα άλλο κομμάτι από το ίδιο περιοδικό, η ιδέα ενό προπολογισμού για την ε, Ευρωζώνη σημαίνει ότι υπάρχει ομοφωνία, ότι προωθείται ομοφωνία για θέματα που δεν προωθούν τη συζήτηση για τον προορισμό 14-20. Ακόμη και οι χώρες που είναι κατά μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων, η ιδέα αυτή αρχίζει να γίνεται όλο και πιο αποδεκτή, εφόσον θα σημάνει αύξηση των εσόδων. Ο Πολωνός υπουργό Εξωτερικών είπε σε μια πολωνική εφημερίδα ότι δεν φοβάται τον προπολογισμό της Ευρωζώνης γιατί ήταν χωριστός από τον γενικό προπολογισμό. Δεν μιλάμε για κάτι που θα γίνει την 1η Ιανουαρίου 2013, Άρα στόχος, ο στόχος αυτός δεν είναι ακόμη αρκετά όριμος. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένας τέτοιος προπολογισμός θα μπορούσε να αρχίσει να ισχύει από το 2014. Και σημείωσε ότι δεν υπάρχει σαφήνεια για το πώς θα χρησιμοποιόταν αυτός ο επιπλέον προπολογισμό. Θα έπρεπε κάπως να έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωζώνης. Οι συζητήσεις για το θέμα αυτό δεν θα λήξουν σύντομα. Και ότι είπε ο κύριος Κάμερον τα εξή. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να υπάρξουν δύο ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί. Ένας για το κοινό νόμισμα, διότι θα πρέπει να υποστηρίξουν ένα τον άλλο περισσότερο και ίσως ένα ευρύτερος προϋπολογισμός για όλους τους άλλους. Βλέπουμε λοιπόν τι κίνδυνοι υπάρχουν, τι διακυβεύεται. Εμείς λοιπόν ως Κοινοβούλιο πρέπει οπωσδήποτε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας. Βεβαίως ε, θα πρέπει να είναι πιο ευφυής η χρήση των πόρων, να έχουμε περισσότερους ίδιους πόρους, αλλά όλα αυτά πρέπει να είναι τμήμα ενός ενιαίου ευρωπαϊκού προπολογισμού. Αυτό πρέπει να κάνουμε σαφές, νομίζω, προς όλους σε αυτή τη συγκυρία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Γιάννη Μιούλτα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους εισηγητές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η προσπάθεια αυτή και πρέπει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δύσκολη αυτή στιγμή να καταφέρουμε να δείχνουμε ότι έχουμε μια κοινή θέση απέναντι στο Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συντοπίσουμε ότι ε, δεν πρέπει τώρα να επιμείνουμε σε επιμέρους ε, παρατηρήσεις που ενδεχομένως να μας διχάζουν, αλλά να επιμένουμε σε μια κοινή γραμμή όσον αφορά όλε αυτές τις φήμες που ακούγονται. Φόρος επί των χρηματιστοτικών συναλλαγών σε 11 χώρες που θα χρησιμοποιηθεί ο ξεχωριστός προπολογισμό για την Ευρωζώνη και το καθεξής. Στη φάση αυτή πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μια ξεκάθαρη θέση. Πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά τη συνθήκη εγώ δεν ξέρω ακριβώς πώς, είναι, πώς έχει κατάσταση. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας και βάσει του δικαιώματο αυτού, στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζουν. Ποια θα είναι λοιπόν η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για όλες αυτές τις ενδιαφέρουσε προτάσεις που ακούγονται για ξεχωριστού προπολογισμού κτλ. Νομίζω ότι στις 26-27 Νοεμβρίου το Συμβούλιο μπορεί να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σίγουρα, αλλά δεν νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να διαπραγματευτούμε βάσει αυτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφανθεί. Αυτή έχει το δικαίωμα πρωτοβουλίας και νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον στο μέλλον να έχουμε μία πάρα πολύ καλή νομική νομοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι λέει η συνθήκη για όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιούτα Χάουγκιν. Ζήτησα τον λόγο για ένα πολύ μικρό τμήμα του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Φυσικά συμφωνώ με αυτά που είπαν και έκαναν ο Ράινερ και ο Ιβάιλο. Σε αυτή την ενδιάμεση έκθεση έχουμε την ίδια δυσχέρεια που για μένα τουλάχιστον είχα και με την έκθεση του Τζοβάνι. Πρόκειται για τους οργανισμούς. Ενδιαφέρουμε για τους οργανισμούς. Δεν είναι ενδιαφέρον της ομάδας μου. Νομίζω ότι είναι κάτι που ενδιαφέρει όλες τις ομάδες. Είναι ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου. Εδώ και τρία χρόνια, εδώ και πάνω από τρία χρόνια, εργαστήκαμε ως διοργανική ομάδα εργασίας και επιτύχαμε ένα αποτέλεσμα που υπεγράφει τον ε, περασμένο Ιούλιο και τώρα υποβάλλονται τροπολογίες και μετά γίνονται συμβασμού, συμβασμοί που τα νερώνουν όλα αυτά. Δεν είναι δυνατόν. Υπήρξε μια διοργανική ομάδα εργασίας, συμμετείχαν όλες ή σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες, συνεργαστήκαμε είχαμε τρία μέλη της Επιτροπής μας, Αν Γένζεν, Κρέσλε και εγώ. Όλοι οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν. Δεν τα κάναμε κρυφά. Δεν συζητήσαμε, αλλά ενημερώσαμε και τους πάντες. Γιατί λοιπόν υποβάλλονται τροπολογίες που έχουν ως αποτέλεσμα να μας κάνουν να νομίζετε ότι ε, οι οργανισμοί αυτοί είναι κάτι εντελώ καινούριο για το οποίο δεν έχετε ακούσει ποτέ τίποτα. Σας παρακαλώ, διαβάστε την κοινή προσέγγιση και διαβάστε και αυτά που συμφωνήσαμε με την Επιτροπή ότι μέχρι τέλους του χρόνου δυστυχώς δεν είναι παρούσα η Μόνικα η ομιλία μου ήταν 50% για την Μόνικα Χολμάγερ Α, ούτε ο κύριο Γκερμπράντι. Αλλά θα πρέπει να το ξαναπώ και αυτού. Σας παρακαλώ, διαβάστε τι συμφωνήσαμε. Αυτά τα οποία συμφωνήσαμε, η Κομισιόν, μετά από αυτά που συμφωνήσαμε, μας δίνει αντικειμενικά κριτήρια και ξέρετε ότι είμαστε μόνο ένα τμήμα της νομοθετικής διαδικασίας. Μα δίνει λοιπόν τα κριτήρια ούτως ώστε εμεί και το Συμβούλιο είτε να κλείσουμε οργανισμούς είτε να συγχωνεύσουμε τέτοιους οργανισμούς ούτω ώστε οι χρηματοδοτήσεις μας να είναι πιο αποτελεσματικές. Αλλά σας παρακαλώ όλα όσα είναι σε αυτό το κείμενο, σε αυτή την κοινή προσέγγιση, σας παρακαλώ αφήστε μας να τα εφαρμόσουμε και τώρα αναφέρομαι στον προπολογισμό 21. Σας παρακαλώ να μας αφήσετε να συνεχίσουμε την εργασία μας Με συγχωρείτε που μίλησα τόσο πολύ. Θα ήθελα να τα πω πριν την ψηφοφορία για την έκθεση του Τζοβάνι, αλλά δεν είχα την ευκαιρία. Δεν χρειάζεται κάθε φορά που επαναρχόμαστε στο θέμα αυτό να θέτουμε να αμφιβόλο όλα όσα επιτύχαμε ενώπιον του Συμβουλίου, έναντι του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να τα αμφισβητούμε και να χρειάζεται να ξαναξεκινάμε από την αρχή. 20, 20, 20 ήταν. Προηγουμένως τώρα είναι 21. Δεν ξέρω τώρα. Δεν πρόλαβα να κοιτάξω. αν θα έπρεπε να υποθεί κάτι για τους οργανισμούς αυτούς, τότε σας παρακαλώ βασιστείτε και αναφερθείτε στην κοινή μας προσέγγιση. Κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να υποθεί τίποτα άλλο. Με συγχωρείτε. Σε ευχαριστούμε Γιούτα. Πολλοί συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στους τονιστές και μετά στους άλλους συναδέλφους. Ο Γκόραν Φέρμ το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ πολύ θερμά τους συνεισηγητές. Έχουν κάνει πραγματικά μια καταπληκτική εργασία και είναι πραγματικά πάρα πολύ θετικό να έχουμε συνεισηγητές για αυτές τις εκθέσεις, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να έχουμε μια μεγάλη ενότητα που είναι πάρα πολύ σημαντικό αν πραγματικά θέλουμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις αυτές. Πιέζονται τώρα ιδιαίτερα τα κράτη-μέλη για να καταλήξουν και αυτά σε μια κοινή θέση πριν το Συμβούλιο που θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο. Ελπίζω βέβαια ότι ε, η χρονική αυτή πίεση δεν θα οδηγήσει στο χειρότερο δυνατό σενάριο που θα έχουμε τελικά κάποια κράτη-μέλη τα οποία θα είναι υπέρ της περικοπής του προπολογισμού αλλά θα είναι υπέρ της ε, ε, κοινής, συγκεκριμένων κοινών πολιτικών αλλά πάλι θα θέλουν μια αύξηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφύγουμε κάτι τέτοιο, γιατί αυτό θα ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο. Τρεις παρατηρήσεις να κάνω. Πρώτον, όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Ξέρω ότι έχουν ε, υποβληθεί συγκεκριμένες τροπολογίες ακόμα και από την πολιτική μου ομάδα. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε εδώ την διατύπωση που είχαμε από την έκθεση ΣΟΥΡ όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική συζήτησα με τους συνηγητές καθώς επίσης και με τον Τζοβάνι Λαβία και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη διατύπωση που είχαμε στην έκθεση της Επιτροπής Σούρα γιατί διαφορετικά θα δημιουργηθούν πραγματικά προβλήματα όσον αφορά την χρηματοδότηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Δεύτερον, Είμαι εισηγητή όσον αφορά το μηχανισμό συνδέοντα την Ευρώπη. Συμβαστική παριθμών 8 από του εισηγητέ έρχεται κάπω σε αντίθεση σε σχέση με τη γνωμοδότηση που έχουμε εγκρίνει στην Επιτροπή Προπολογισμών. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο βέβαια γίνεται κάτι τέτοιο. Λέγεται τουλάχιστον κατά τη διάρκεια τα πρώτα χρόνια θα πρέπει να σεβαστούμε την εθνική κατανομή πόρων στα πλαίσια του Ταμείου αυτού. Να σα πεθυμίσω όμω ότι ο στόχο τη πρόταση είναι να καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να καταλήξουμε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο και σιγά σιγά να απομακρυνθούμε από την εθνική χρηματοδότηση και την εθνική κατανομή πόρων. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο θέλουν να διατηρήσουν την διατύπωση αυτή οι συνεισηγητέ, αλλά μην πάμε παραπέρα γιατί θα χάσουμε ουσιαστικά τους βασικούς στόχου και την προστιθέμενη αξία του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη. Μπορώ να σεβαστώ την διατύπωση αυτή, αλλά ας μην πάμε παραπέρα. Και κάτι τελευταίο, το βασικό ζήτημα, συζήτηση του προπολογισμού για την Ευρωζώνη και το καθεξής. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μείνουμε στι αρχές μας δηλαδή στην τροπολογία τη δικιά μου την 175, καθώς επίσης και στην τροπολογία κάλφιν παριθμό 15. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κανένα λόγο να απομακρυνθούμε από τη βασική μας θέση αρχής όσον αφορά την ενότητα και την καθολικότητα του κοινοτικού προπολογισμού. Ξέρω ότι διεξάγεται αυτή τη στιγμή μια συζήτηση, ξέρω ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυ στη συζήτηση αυτή, αλλά φοβάμαι πολύ ότι αν αποδεχθούμε οτιδήποτε άλλο αυτή τη στιγμή, τότε ουσιαστικά θα καταλήξουμε πολύ γρήγορα σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Α μην αναλύουμε αυτή τη στιγμή τι λέει, τι κάνει ο κύριο Κάμερον. Νομίζω ότι είναι σαφέ ότι ακόμα και αν μπορεί να δώσει κάποιε θετικέ εξηγήσει για τι προσδοκίε του, όσον αφορά τον ξεχωριστό προπολογισμό, ξέρετε ότι από την άλλη αυτό που θέλει να πετύχει είναι μείωση τη συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτό είναι σαφέ. Αν ακολουθήσουμε λοιπόν το συλλογισμό του, φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε σε τεράστια προβλήματα. Σαφώς θα πρέπει να παρακολουθήσουμε βέβαια τις όλες εξελίξεις. Ξέρω τα πράγματα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Θα μπορούσαμε δεχομένως κάπως να συντονιστούμε μεταξύ ημών προτού την τελική προθεσμία που έχουμε για την Ολομέλεια. Να δούμε δηλαδή αν έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο σε μια συνεδρίαση συντονιστών, σε μια συνάντηση με τους εισηγητές θα μπορούσαμε να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις προτού αποφασίσουμε οριστικά για το πώς θα πρέπει να ψηφίσουμε κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας. Μέχρι στιγμής πάντως τίποτα δεν με έχει πείσει ότι θα πρέπει να κάνουμε τίποτα περαιτέρω από το να παραμείνουμε σε αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε Γκέραν, ο κύριος Κλούτεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία επίκριση. Δεν με καλέσατε στις διαπραγματεύσεις για τον συμβασμό. Δεν είδα εδώ κανένα email. Καλό θα ήταν να μας είχατε καλέσει. Στις άλλες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, πάντα προσκαλούμεθα για το περιεχόμενο. Μπορώ να υποστηρίξω πολλά από αυτά και θα υποστηρίξουμε αυτά που υπόθηκαν για τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε όλες τις πολιτικές ομάδες γι' αυτό. Και τα είπα και στην ομάδα επαφών αυτά. Αλλά είναι σημαντικό να μας ε, προσκαλείτε στις διαπραγματεύσεις για τις συμβαστικές τροπολογίες. Για το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που αναφέρεται, θέλω να πω κάτι στην έκθεση, θα ήταν σκόπιμο, κατά τη γνώμη μας, ως ομάδα, να το πούμε σαφέστερα κάπως. Στην ΕΚΟΝ το συζητάμε πολύ συγκεκριμένα αυτό το θέμα αυτό. Η ΕΚΟΝ ε, θεωρεί με ευρία πλειοψηφία ότι θα έπρεπε να εισαχθεί αυτός ο φόρος. Πιστεύω λοιπόν ότι και εδώ θα έπρεπε να υποθεί σαφέστερα να τονιστεί περισσότερο. Ένα θέμα για το οποίο μπορούν να συνεργαστούν διάφορες επιτροπές. Αναφέρεται είπα, αλλά να τονιστεί περισσότερο. Και για λόγους πολιτικής έναντι των χρηματαγορών, να αναφέρουμε ότι είναι μια δυνατότητα για να ενισχύσουμε τους ίδιους πόρους. Θα ήθελα λοιπόν να υποθεί σαφέστερα. Σας ευχαριστούμε. Συντόνια. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όλους όσοι ευχαρίστησαν τους εισηγητές, καθώς επίσης και τους βοηθούς τους, προκειμένου να καταλήξουν σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες που θεωρώ ότι αντικατοπτρίζουν τις συζητήσεις που ήδη είχαμε εδώ και θεωρώ ότι αποτελούν μια πολύ καλή βάση προκειμένου να καταλήξουμε σε μια ψηφοφορία αύριο. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τρία ζητήματα. Τις συμβαστικές τροπολογίες, τις τροπολογίες που μείναν εκτός και που πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε ενδεχομένω και τρίτον να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την δυνατότητα πιθανής δημιουργίας ενός προπολογισμού για την Ευρωζώνη. Όσον αφορά τους συμβιβασμού, θεωρώ ότι είναι πολύ λογική, συμπεριλαμβάνουν πολλές τροπολογίες, είναι σωστή. Θα μπορούσα να επικεντρωθώ σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες με τις οποίες δεν συμφωνώ. Αποτελούν εξαίρεση βασικά. Το βασικό ζήτημα έχει να κάνει με την κλιματική πολιτική, την πολιτική για τις κλιματικές αλλαγές. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στη συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 6 Δεν μπορώ να συμφωνήσω με μία δήλωση που γίνεται σε αυτήν τη συμβαστική τροπολογία και που έχει να κάνει με την συμπερίληψη μέτρων για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών τουλάχιστον σε ένα 20% των μέτρων που προβλέπονται στον κοινοτικό προπολογισμό για τις κλιματικές αλλαγές. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό να αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα ποσοστό 20%, ιδιαίτερα υψηλό. Ενδεχομένως βέβαια να μου διαφεύγει κάτι το οποίο πρώτερα συμφωνήσαμε, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει μια τόσο απόλυτη δήλωση στο παρελθόν. Ενδεχομένως να μπορούμε να το διευκρινίσουμε βέβαια αυτό λίγο αργότερα. Συμφωνώ έπειτα με όλους τους υπόλοιπους συμβιασμούς. Έρχομαι στο συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 11. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να Βλέπουμε εδώ πέρα τις άμεσες πληρωμές ε, στους ε, αγρότες, καθώς επίσης και τα κονδύλια τα οποία προέρχονται από το Αγροτικό Ταμείο στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Δεν θα ήταν καλό να έχουμε σε μία δήλωση και αυτά τα δύο είδη πόρων. Ενδεχομένω να πρέπει να επεξεργαστούμε τη συμβαστική αυτή τροπολογία ή να τη χωρίσουμε σε δύο τμήματα άμεσες πληρωμές και ανάπτυξη της υπαίθρου δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τουλάχιστον στο πλαίσιο αυτό της συμβαστικής τροπολογίας. Μία άλλη παρατήρηση πάλι για τους συμβασμούς. Μάλλον ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Να επανέλθω τώρα σε κάποιες μονομένες τροπολογίες. Εγώ ίδια αλλά και άλλοι συνάδελφοι είχαμε υποβάλει κάποιες τροπολογίες που είχαν να κάνουν με το ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει μια διάσταση του προπολογισμού υπέρ της ανάπτυξης και νομίζω ότι ε, πολλοί έχουν ταχθεί κατά κάτι τέτοιο πρόσφατα. Υπάρχουν δηλαδή πολλά επιχειρήματα που ε, θέτουν ένα αμφιβόλο το αν τελικά ο κοινοτικό προπολογισμό είναι υπέρ τη οικονομική ανάπτυξη, υπέρ τη δημιουργία θέσεων εργασία, αν πραγματικά οδηγεί σε περισσότερε επενδύσει. Εγώ πιστεύω ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα ζητούσα λοιπόν από τους εισηγητές να επανεξετάσουν τις τροπολογίες αυτές οι οποίες υπογραμμίζουν το ρόλο αυτό του κοινοτικού προπολογισμού, το ότι προωθεί δηλαδή την οικονομική ανάπτυξη και ότι δημιουργεί τελικά θέσεις εργασίας. Κάτι όσον αφορά τώρα τον προπολογισμό της Ευρωζώνης, τον λεγόμενο προπολογισμό της Ευρωζώνης. Λοιπόν, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι συμβαίνουν διάφορα πράγματα αυτή τη στιγμή. Παράλληλα, δεν έχουμε λάβει αρκετές πληροφορίες ακόμα δεν εμπλεκόμαστε εμείς δυστυχώς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτές τις ενεξελίξει προετοιμασίες στην δημιουργία, αν μπορούμε να την αποκαλύσουμε έτσι, ενός προπολογισμού για την Ευρωζώνη. Υπάρχουν λοιπόν πολλά εκκρεμή ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Επομένω, η ερώτησή μου είναι καταρχάς, εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώ θα καταφέρουμε να συμμετάσχουμε στην θεωρητική αυτή καζόμενη δημιουργία ενός προπολογισμού για την Ευρωζώνη. Για μένα αυτό παραμένει ακόμα σαφές και ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι είμαστε απλοί παρατηρητές των όσων περιγράφουν ε, οι εφημερίδες και άλλα μέσα. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, κατά την άποψή μου, το ελάχιστο το οποίο επιβάλλεται να κάνουμε είναι να ζητήσουμε να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να υπάρχει δηλαδή μια κοινοβουλευτική διαδικασία σε σχέση με τις εξελίξεις αυτές. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες των συναδέλφων που έχουν να κάνουν με την απουσία κάποια ενημέρωση ή την έλλειψη δηλώσεων εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάτι τέτοιο πρέπει να απαιτήσουμε. Να δούμε δηλαδή ποια είναι η θέση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να έχει κάνει κάποια δήλωση, να κάνει κάποια δήλωση η σε περίπτωση που δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Και κάτι ακόμα. Επί του παρόντος δεν θα ήθελα να καταλήξουμε σε μία ξεκάθαρη οριστική τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο ακόμα επί του ζητήματος αυτού. Δεν νομίζω ότι στα πλαίσια της ε, ενδιάμεσης έκθεσης των εισηγητών Μπέγκε και Κάλφιν να μπορούμε να συμπεριλάβουμε και μία άποψή μας όσον αφορά τον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Είναι πάρα πολύ νωρίς, πρέπει να επιληφθούμε ακόμα περισσότερο του στήματος αυτού. Εν γέννη πιστεύω ότι στην έκθεση αυτή θα πρέπει να μείνουμε σε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Νοεμβρίου, καθώς επίσης και το Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Και θα πρέπει να κάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μπλακούμε και εμείς στην, στον προπολογισμό της Ευρωζώνης. Ευχαριστούμε την συντονία. Ο κύριος Ναράν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λίγο χρόνο θα πανίσω γιατί πολλά ακούστηκαν, προακούστηκαν που είναι άκρος ενδιαφέροντα και με βρίσκουν ως επιτοπλίστων σύμφωνο. Συμφωνώ με τον Γκόραν Φέρμα και τον Ράιτμαρ σε σχέση με τις πρωτοβουλίες από κυβερνητικής πλευράς ιδιαίτερα για να δούμε κατά πόσο θα υπάρξει ένας ξεχωριστός προϋπολογισμός για την Ευρωζώνη και τι θα γίνει με το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μέσα στα πλαίσια και της αντιμετώπισης του ΦΠΑ. Είναι ιδιαίτερα η αγωνιώδης η κατάσταση που γνωρίζουμε στο παρόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές καταρχήν και καταλαβαίνω το ότι να υφάνουμε συμβιβασμούς είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο. Ως προς το συμβασμό 10 που αναφέρεται στην παράγραφο 21 που αρχικά μιλούσαμε για για μια περίοδο, για ένα επίπεδο που αφορά την περίοδο 2007-2013, νομίζω ότι ε, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Ε, αναφερόταν θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στο επίπεδο της περίοδου 7-13. Νομίζω λοιπόν ότι δεν αρμόζει σε αυτή την έκθεση αυτού του τύπου οι αναφορές. Μιλάμε για περικοπές μέσα στα πλαίσια μίας δημοσιονομικής λιτότητας, κάτι το οποίο αποδυναμώνει την έκθεση συνολικά. Θα ήθελα η έκθεση να είναι μία στεναρή έκθεση με την ευρύτατη, ευρύτερη δυνατή συνένεση. Και αυτό θα ήθελα να το εντάξω στην εργασία των εξαιρετικών μας συντακτών. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να τονίσω ότι ως προς την παράγραφο 21 δεν ε, ε, είμαι σύμφωνος ως προς την αρχική διατύπωση. Ναντέσνα Σίνσκι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τους εισηγητές για την εξαιρετική αυτή έκθεση ε, και αυτό το θαραλέο βήμα και διάβημα για αυτή τη μεγάλη αλλαγή ως προς τις άμεσες πληρωμές και τους συμβιβασμούς που βρήκαμε γενικότερα. Και ως προς τον αγροτικό τομέα, φτάσαμε σε συμφωνίες, σε μια συμφωνία για την Βουλγαρία, για την αντιμετώπιση των αγροτών μέσα στα πλαίσια αυτού του συμβιβασμού θα πρέπει οι άμεσες πληρωμές να είναι ίσες και δίκαιες σε σχέση με τις άλλες πληρωμές. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τους εισηγητές για αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε Ναντέζνα. Ο κύριος Κουντμάνης. Θα ήθελα να υποστηρίξω τους εισηγητές για τους δύο συμβασμούς στην παράγραφο 21, 10 και 11. Τους συμβιβασμούς 10 και 11, επί της παραγράφου 21. Δεν νομίζω ότι έχουν γίνει και πολλά, αλλά θα τους υποστηρίξω αυτούς τους συμβιβασμούς παρόλο που δεν καλύπτομαι απόλυτα. Πολύ καλή θέση και θα υπερψηφίσω αύριο. Τζοβάνι Λαβία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους εισηγητές για την εξαιρετική τους εργασία και θα ήθελα να σταθώ στο συμβιβασμό 11 που σχετίζεται με την ΚΑΠ. Εγώ είχα υποβάλει και ορισμένες τροπολογίες πιο ριζοσπαστικές για την ΚΑΠ σε σχέση με το συμβασμό αυτό. Θα ήθελα όμως να τονίσω δύο πτυχές. Υπάρχει μια σειρά τροπολογιών που αναφέρεται στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε όχι μόνο στο πάγωμα του προϋπολισμού του 2013, αλλά στις οροφές σε σχέση με το προηγούμενο MFF. Θα ήθελα, λοιπόν, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την οροφή δαπανών σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό, όπως αντιμετωπίζεται φέτος. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και ορισμένες τροπολογίες των σοσιαλιστών για μια καλύτερη διασαφήνιση. Ως προς το πρώτο και δεύτερο πυλώνα, ο συσχετισμός δεν είναι σωστός, διότι πολλές φορές έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα ο πρώτος με το δεύτερο πυλώνα. Και γι' αυτό νομίζω ότι η ενιαία βάση είναι σωστή. Το τρίτο θέμα αφορά τις ενυπάρχουσες διαφορές μεταξύ κρατών, περιφερειών και αγροτών. Γιατί στην πρόταση της Επιτροπής, όπως θα θυμόσαστε, υπήρχε η πρόταση μείωσης κατά εν τρίτον. Τώρα στη συζήτηση της Επιτροπής Γεωργίας μιλάμε για μειώσεις. Στην πρόταση συμβιβασμού μιλάμε για συρρήκνωση, μείωση του χάσματος. Νομίζω ότι αυτό συμβαδίζει με την, επίτρο... με την πρόταση της Επιτροπής και την πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας. Θα πρέπει να μιλήσουμε για, όχι για closing up, αλλά reducing, κάπως να, να εντάξουμε τη λέξη της μείωσης του, του περιορισμού αυτού του χάσματος. Ευχαριστούμε κύριε Λαβία. Η Ίγκε Χέσλε. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ήταν η κατάσταση μέχρι τώρα για το πολιτέ πλαίσιο και αυτή η ανακοίνωση ενό προπολογισμού τη Ευρωζώνη μα πέφτει στο κεφάλι. Το θέμα είναι πώ θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Τι θα είναι αυτό το προπολογισμό τη Ευρωζώνη. Δεν καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω πώς ε, θα διατυπωθεί Ποιοι θα αποφασίσουν επίσης. Θα αποφασίσουν αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων όπως προηγουμένως οι βασιλείς στα μοναρχιά καθεστώτα μόνοι τους. Με τι διαδικασία θα υπάρξει απόφαση. Θα υπάρξουν αποφάσεις των εθνικών κοινοβουλίων. Όποιος ε, είχε αυτή την ιδέα και μας την είπε, μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Οι Βρετανοί, συμφωνώ με τον Γκέραν, έχουν κάθε λόγο να την υποστηρίξουν και πρέπει οπωσδήποτε να αντιπαρατεθούμε με αυτή την ιδέα. Το κοινοβούλιο μας πάντα έβρισκε τρόπους να αποφασίζει για τα θέματα του ευρώ. Το Συμβούλιο δημιουργεί το πρόβλημα. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να, να αντιτεθούμε σε αυτές τις ιδέες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους εισηγητές ε, για την ε, ποιοτική τους εργασία και τη διαθεσιμότητά τους, η οποία ποτέ δεν διαψεύστηκε. Πριν μιλήσω ως σοσιαλιστής θα ήθελα να επανέλθω σε δύο παρεμβάσεις, ε, Φέρμ και Γιούτα Χάουκ, για να πω ότι ως προς το συμβιβασμό 8 που αφορά τη δυσκολία που έχουμε με τα 10 δις του Connecting for Europe. Θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για αυτό το μέσον μεταξύ της Επιτροπής Μεταφορών και Ρέτζι και των χωρών συνοχής που έχουν βεβαίως μεγάλες ανησυχίες. Θα ήθελα να πω στον ε, Γκέραν ότι αυτή είναι μία μαξιμαλιστική προσέγγιση αν δεν είχαμε αυτό το at least, αυτό το at least οφείλω να πω ότι με ενοχλεί κάπως αυτό το, αυτή η μνήα του τουλάχιστον. Δεύτερον, συμμερίζομαι τα σχόλια της Γιούτα σε σχέση με την τροπολογία 21. Είχαμε φτάσει σε μια συμφωνία και είναι σαν να την αμφισβητούμε. Βεβαίως υπάρχει μια δημοσιονομική προσέγγιση, θέλουμε βελτιστοποίηση, ε, ένα συντονισμό, αλλά αναρωτιέμαι κατά πόσο πίσω από αυτό κρύβονται άλλα, παρόλο που έγιναν από την ομάδα μου και από την αντιπροσωπεία μου. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει κυβερνητικός δάκτυλος εδώ, αυτών που δεν θέλουν ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θέλουν να χάσουμε μέσα ολοκλήρωσης. Άρα είμαι κάπως επιφυλακτικός ως προς το Σύμβασμο 21. Όσον αφορά το προϋπολογισμό της Ευρωζώνης, αυτό αποτελεί αδυσόπιτη εξέλιξη των καιρών. Όταν αρχίσαμε με την ε, αγορά είπαμε ότι θα προωθήσουμε το κοινό νόμισμα. Πολλοί μείναν εκτός και δεν μπορεί παρά να υπάρχει και νομισματική αλληλεγγύη. Και όλες, όλα αυτά ε, τα οποία βρίσκονταν σε λανθάνουσα μορφή βγαίνουν στην επιφάνεια. Εδώ μιλώ και για, τον, και για το τραπεζικό πακέτο και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε τον προεπολισμό της Ευρωζώνης εάν ανακύψει θα υπάρχει η ίδια διαχείριση με τον γενικό προεπλασμό. Τι θα γίνει όμως ε, με αυτούς που διάλεξαν το opt-out που θα συνεισφέρουν ε, όλο ένα και λιγότερο. Δηλαδή τι θα γίνει με αυτό το υπόλοιμα προϋπολογισμού αν όλοι ζητήσουν ρήτρα αυτοεξαίρεσης. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί δεν πρόκειται για επιφαινόμενο, πρόκειται για μία ε, αδυσόπιτη εξέλιξη και θα υπάρξουν και συγκεκριμένες συνέπειες του προϋπολογισμού αν δεν υπάρχει μια συνεπής νομισματική πολιτική. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Πολύ ενδιαφέρουσα και πλούσια συζήτηση που είχαμε και καλύψαμε όλες τις πτυχές των προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Εναπόκειται πάλι βέβαια στους συνεισηγητές μας να τους ευχαριστήσουμε για την πολύ καλή δουλειά που κάνανε, μια ομαδική συλλογική εργασία και λάβαν υπόψη τους τι παρατηρήσει πολλών συναδέλφων. Να κάνω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχά, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω, όπω το έκανε και ο Ράιμερ, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε μπροστά μα, το οποίο είναι πάρα πολύ πιεστικό. Θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Υπάρχουν πολλέ μάλλον εκθέσει. Το σύνολο πάντως του πακέτου MFF θα το ψηφίσουμε αύριο λαμβάνω υπόψη τις παρατηρήσεις σας ότι έχετε ακόμα κάποιες ενστάσεις και συγκεκριμένε τροπολογίες ή συμβαστικές τροπολογίες που πρέπει να διευκρινίσουμε. Την επόμενη τώρα εβδομάδα μετά την ψηφοφορία που θα έχουμε, για την προσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή της Επιτροπής των Προπολογισμών, οι εισηγητές και εγώ, θα συναντηθούμε στο Λουξεμβούργο με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων μας κάλεσαν να συμμετάσχουμε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων δεν θα συναντήσουμε απλώς δηλαδή την Κυπριακή Προεδρία αλλά το σύνολο των Υπουργών όπου θα έχουμε ένα γεύμα εργασίας αφιερωμένο στο ζήτημα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Η ψηφοφορία λοιπόν που θα έχουμε αύριο θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Βέβαια, δεν είναι η τελική οριστική ψηφοφορία της Ολομέλειας, αλλά ξέρετε ότι γενικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλους ε, ανάλογους οργανισμούς, πολύ συχνά η ψηφοφορία σε μια Επιτροπή Προπολογισμών με τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια ουσιαστικά ταυτίζονται συνήθως. Πρώτη παρατήρηση αυτή. Δεύτερον, Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο για να χαρούμε τελικά κιόλας για την πολιτική επιτυχία που είχαμε, επιβάλλοντας τη συζήτηση αυτή όσον αφορά το τμήμα που αφορά τους πόρους του προπολογισμού. Από ό,τι φαίνεται τελικά αντιστρέφουμε το βάρος απόδειξης αυτή τη στιγμή. Θα θυμάστε ότι στην Επιτροπή μας αυτή, στην Επιτροπή των Προπολογισμών, ήμασταν οι πρώτοι που είχαμε πει ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο έτσι, δεν μπορούμε να χρηματοδοτούμε κατά αυτόν τον τρόπο τις αρμοδιότητες και τις νέες αρμοδιότητες που προκύπτουν από τη συνθήκες της Λισαβόνας, αν πραγματικά μείνουμε κλεισμένοι σε ένα πάρα πολύ περιοριστικό σύστημα το οποίο προβλέπει χρηματοδότηση μόνο από τα κράτη-μέλη, από τους εθνικούς προπολογισμούς το σύστημα δεν ήταν καλό πριν την κρίση, έχει επιδεινωθεί τώρα με την κρίση. Αρχίσαμε λοιπόν να μιλάμε για το πρόβλημα αυτό και τότε σε μία πρώτη φάση είχαμε πάρα πολλές αντιδράσεις εκτός Κοινοβουλίου. Απόλυτο σκεπτικισμός, ηρωνικά σχόλια. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι του 2011, όταν ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι είχε τότε ξεκινήσει εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμερίζεται κάπως τη δική μας την ανάλυση, έδωσε μια συνέντευξη τον Αύγουστο για το ζήτημα αυτό και είχε προκαλέσει τεράστια αναστάτωση και αντίδραση σε όλα τα Υπουργεία Οικονομικών. Σήμερα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις επιτάπητος και εν τέλει τελικά κανείς δεν διαφωνεί ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το κεφάλαιο των πόρων. Δίστανται σίγουρα πάρα πολύ απόψε όσον αφορά το περιεχόμενο του στόχου αυτού. Πάντως αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι ε, αρχίζει να στρέφεται η κοινή γνώμη περισσότερο προς εμάς, απέναντι σε αυτούς, σε αντίθεση με αυτούς που θέλουν να διατηρήσουν την υφιστάμενη κατάσταση, το status quo. και είχαμε κάνει και συγκεκριμένε προτάσει ψηφίζοντα τον προπολογισμό του 2011 και τότε είχαμε προναφερθεί επίση και στο φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όλα αυτά αποτελούν απόδειξη του γεγονότο ότι όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίζει να ασχολείται πραγματικά με ένα ζήτημα, εμένει σε ένα ζήτημα και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό, τότε πραγματικά σημειώνεται πρόοδος από την αρχή της όλης ιστορίας όσον αφορά τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών υπήρχε μια κάποια αμφισημία. Υπήρχε ή το σενάριο Λεβαντόφσκι και το σενάριο Σεμέτα. Ο Σεμέτα μας πρότεινε να υπάρχει ο φόρος αυτός χωρίς να υπάρχει διασύνδεση με τον προπολογισμό. Ο Λεβαντόφσκι με τη σειρά του είπε ότι εφόσον δημιουργηθεί ο φόρος αυτός θα πρέπει να αποτελέσει ίδιο πόρο. Και τι βλέπουμε σήμερα. Ήδη από χθε ουσιαστικά έχουμε την εξή κατάσταση. Υπάρχουν πλέον οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να έχουμε μια ενισχυμένη συνεργασία. Και διάμεσα πετύχαμε μία ακόμα επιτυχία, αρχικά σε σχέση με το σχέδιο του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, όπου θα θυμάστε ότι στην αρχή είχαμε διάφορα ερωνικά σχόλια και αντιδράσεις από τα κράτη-μέλη που λέγανε μα ούτως ή άλλως θα χρειαστεί απόλυτη ομοφωνία, κράτη όπως το Λουξεμβούργο, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασιλείο, υποτίθεται δεν θα δέχονταν ποτέ μια τέτοια ιδέα, επομένω είχαν καταδικάσει από την αρχή την ιδέα αυτή. Και τώρα βλέπουμε όμως ότι μπορούμε να έχουμε μία ενισχυμένη συνεργασία. Σίγουρα δεν θα καταφέρουμε να συλλέξουμε τόσους πόρους όσο αν συμμετείχαν και τα 27 κράτη-μέλη, πάντως αυτό που βλέπουμε είναι ότι από νομικής και πολιτικής πλευράς, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, μπορούμε να έχουμε πόρους από τον φόρο αυτό, οι οποίοι θα πάνε στον κοινοτικό προπολογισμό και θα επιτρέψουμε τη σειρά τους να μειωθεί η εθνική συνεισφορά των κρατών μελών προς τον κοινοτικό προπολογισμό. Ήδη από χθε έχουμε περισσότερα από 9 χώρες, 11 πλέον χώρες, που έχουν συνυπογράψει μια πρωτοβουλία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από τη συνθήκη, υποχρεωμένη να θέσει επιτάπητος να κάνει μια πρωτοβουλία όσον αφορά το νομικό μέσο της ενισχυμένης αυτής συνεργασίας. Ενισχυμένη λοιπόν πλειοψηφία απαιτείται πλέον στα πλαίσια του Συμβουλίου προκειμένου να τεθεί ενισχύ, να εγκριθεί αυτή η ενισχυμένη συνεργασία. Το Ηνωμένο Βασίλειο μας είπε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει, αλλά ότι δεν πρόκειται να εμποδίσει και τη διαδικασία. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πλέον πάρα πολύ δυνατό να εγκριθεί και να ελοποιηθεί αυτή η ενισχυμένη συνεργασία. Να δημιουργηθεί λοιπόν η ενισχυμένη αυτή συνεργασία σε συνθήκες όμως πολύ μεγάλης ε, ασάφειας όσον αφορά τη μετέπειτα χρήση που θα γίνει των πόρων αυτών που θα συλλεχθούν. Στα πλαίσια των 27 κρατών μελών, αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες χωρών. Έχουμε τις χώρες αυτές οι οποίες δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν και δεν συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται για τη δημιουργία ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, με την προϋπόθεση όμως να ενισχύει αποκλειστικά τους εθνικούς προπολογισμούς αυτός ο φόρος. Έχετε στη συνέχεια τις χώρες εκείνες που ακολουθούν τη γραμμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή τις χώρες εκείνες που θέλουν ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να χρηματοδοτηθούν όχι αποκλειστικά, αλλά σε ένα πολύ μεγάλο τμήμα, να χρηματοδοτηθεί, με συγχωρείτε, ο κοινοτικό προπολογισμό. Και στη συνέχεια έχουμε και την κατηγορία των χωρών εκείνων που αναμφίβολα, και λέω αναμφίβολα γιατί δεν έγινε καμία επίσημη δήλωση, αλλά παρασκηνιακά λένε και κάνουν πολλά πράγματα. Χώρες λοιπόν οι οποίες αναμφίβολα θα ήταν υπέρ όλο ή μέρο του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτηθεί ένας προϋπολογισμός της Ευρωζώνης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επίσης για να εγγυηθούμε τον ε, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή άλλα τέτοια μέσα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές στάσεις όσον αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το φόρο αυτό. Το καλό νέο τώρα για μας είναι ότι υφίσταται, ότι το σύστημα λειτουργεί, ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία και επομένως μπορούμε πλέον να πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κάτι σε ένα είδος πολιτικής συμφωνίας όσον αφορά την μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων που δεν θα περιορίζεται μόνο στη χρήση του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αλλά που θα περιλαμβάνει σημαντικό του μέρος το φόρο αυτό. Και μία ακόμα παρατήρηση, τελευταία παρατήρηση. Όσον αφορά το σχέδιο αυτό κεντρικού προπολογισμού για την Ευρωζώνη. Πρόκειται για μία ιδέα που δημοσίως για πρώτη φορά φάνηκε σε ένα έγγραφο, πολύ σύντομα, ένα έγγραφο του ίδιου του Προέδρου Φαν Ρομπόι. Πολλοί τότε είπαν ότι ας μην βρεθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτελεσμένου, πώς είναι ποτέ δυνατό να υπάρχει ένα τέτοιο έγγραφο χωρίς να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να εμποδίσουμε ούτε τις κυβερνήσεις, ούτε τον κύριο Φαν Ρομπόη να κάνει τέτοιες δηλώσεις ή να συντάσει τέτοια έγγραφα, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι για μία ακόμη φορά οι πραγματικές αποφάσεις προσανατολισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής δεν λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά από το Συμβούλιο και από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και αυτό με τη σειρά του δημιουργεί ένα θεμελιώδες πρόβλημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρα από τις νομοθετικές αρμοδιότητες που έχουμε από νομικής πλευράς, πώς μπορούμε να αυξήσουμε και την πολιτική μας επιρροή στα πλαίσια του θεσμικού αυτού οργάνου που λαμβάνονται πραγματικά οι αποφάσεις και το οποίο δεν είναι πλέον το Συμβούλιο των Υπουργών. Ενδεχομένω να πρέπει και στο μέλλον να επανασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Ενδεχομένω να πρέπει να συζητήσουμε και με του συναδέλφου από την Επιτροπή Σταγματικών Θεμάτων. Το ζήτημα αυτό δεν άπτεται μόνο του προπολογισμού. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα ζητήματα που θα πρέπει να μα απασχολήσουν σε αυτό το πλαίσιο, όπω για παράδειγμα η δημιουργία τη Τραπεζική Ένωση. Και η δημιουργία τη Ένωση αυτή θέτει τα ζητήματα αυτά συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που βλέπουμε ξεκάθαρα πάντω είναι ότι η ιδέα αυτή δεν είναι απλώς μια φάνταστη ιδέα του Προέδρου Φαν Ρομπόη, αλλά ότι πίσω από την ιδέα αυτή ουσιαστικά υπάρχει υποστήριξη ορισμένων κρατών μελών. Κράτη-μέλη τα οποία σκέφτονται ήδη για το ζήτημα αυτό, εργάζονται με αριθμητικά στοιχεία. Και οποιαδήποτε είναι, και είναι η απόψή μα για την ιδέα αυτή, εγώ δεν είμαι εκ των προτέρων εχθρικός, Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι το να αναφερθούμε αυτή τη στιγμή στην ιδέα αυτή είναι ό,τι χειρότερο, είναι η χειρότερη δυνατή στιγμή. Γιατί βρισκόμαστε στη χρονική εκείνη στιγμή που θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για τα αριθμητικά στοιχεία του προπολογισμού για την περίοδο 2014-2020. Αν αρχίσουμε να μιλάμε και για αυτό το θέμα τώρα, θα καταστήσουμε τις διαπραγματεύσεις ακόμα πιο δύσκολες. Και ουσιαστικά θα συμβάλλουμε μόνο στο να δημιουργηθεί πολύ μεγαλύτερη σύγχυση. Γιατί πέρα από την ε, ιδέα για τον προπολογισμό της Ευρωζώνης τίθενται και άλλα ζητήματα. Τα ζητήματα τα οποία ανέφεραν οι συγητές και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Πρώτον, ποια θα είναι η χρηματοδότηση ενός τέτοιου προπολογισμού. Εγώ πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Μου κάνει εντύπωση να ακούω χώρες που ανήκουν στην περίφημη λέσχη του better spending, των καλύτερων δαπανών, που θέλουν ουσιαστικά να υπάρχει μία μείωση 100 δισεκατομμυρίων σε σχέση με την πρόταση για το κοινοτικό προπολογισμό. Θέλουν να μειώσουν τη δικιά τους την εθνική συνεισφορά και από την άλλη λένε ότι θέλουν να δημιουργήσουν έναν νέο προπολογισμό για την Ευρωζώνη που θα τους επιβάλλει μια νέα εισφορά πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως πώς θα γίνει κάτι τέτοιο. Πώς θα χρηματοδοτηθεί ένας τέτοιος προπολογισμός, από τους εθνικούς προπολογισμούς, από τους ιδίους πόρους μήπως. Μα είναι τα ίδια αυτά τα κράτη τα οποία δεν θέλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ιδίους πόρους. Αν όμω τελικά ο προπολογισμό αυτό δεν του αφορά, αυτό φαίνεται, τότε εκεί δεν έχουν πρόβλημα, δέχονται του ίδιου πόρου, αρκεί να αφορά ένα προπολογισμό τη Ευρωζώνη και όχι ένα προπολογισμό που να του αφορά. Αβεβαιότητα λοιπόν όσον αφορά τη χρηματοδότηση, και ανησυχίε όσον αφορά τη χρηματοδότηση στη συνέχεια, σε τι θα πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο προπολογισμός. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, εξαρτώνται αυτή τη στιγμή από κοινοτικού προπολογισμούς, όπως για παράδειγμα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Κάνουν πάρα πολλές θυσίες αυτές οι χώρες αυτές θα μπορούσαν ουσιαστικά να ενισχυθούν, λένε, μέσω του προπολογισμού αυτού για την Ευρωζώνη. Μα ουσιαστικά είναι σαν να αντικαθιστούμε όλα τα άλλα μέσα τα οποία έχουμε, όπω το Ταμείο Συνοχή ή όλα τα υπόλοιπα ταμεία. Τι θα έχουμε τελικά, μια συνοχή 27 κράτη-μέλη, μια, συνοχή, μια πολιτική συνοχή μόνο για την Ευρωζώνη. Και αναφέρομαι και στις ε, χώρες αυτές οι οποίε δεν βρίσκονται στην Ευρωζώνη, αλλά έχουν καταβάλει και αυτέ φοβερέ θυσίε. Δεν θα καταφέρουν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Αναφέρομαι στην Λετωνία, στη Ρουμανία και σε πολλέ άλλε χώρε. Υπάρχει επίσης ανασφάλεια και ως προς το χρονοδιάγραμμά μας. Δεν πρόκειται για κάτι που θα τεθεί σε εφαρμογή φέτος ή το 2013, αλλά θα ισχύσει αυτό το καθεστώς από το 2014 μαζί με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ποια θα είναι η νομική βάση σε αυτή την περίπτωση. Θα υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία μέσα στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας ή χρειάζεται νέος προϋπολογισμός. Υπάρχει μία σωρία ερωτημάτων. Και θα ήθελα να κάνω την εξής ε, υπόδειξη. Όπως υποδεικνύουν και οι εισηγητές, δεν θα πρέπει εκ των προτέρων να απορρίψουμε αυτό το πλαίσιο. Απλώς θα πρέπει να επεξηγήσουμε στεναρά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ε, αποφανθεί ως προς το MFF αν δεν έχει περισσότερες ε, διευκρινήσεις για τους πολιτικούς στόχους, τη χρηματοδότηση, το περιεχόμενο και το νομικό καθεστώς της Ευρωζώνης και του ενδεχόμενου προϋπολογισμού. Αυτή είναι η δική μου σύσταση. Και αυτό να το πούμε πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Φυσικά, διαφορετικά. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου προχωρήσει αυτό το θέμα, εάν υπάρξει απαρχή συμφωνίας, τότε θα βρεθούμε ενώπιον τετελεσμένου. Εάν λοιπόν έχουμε επιφυλάξει ερωτήματα, νομίζω θα πρέπει να τεθούν πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αύριο δηλαδή αυτό προβλέπεται και στο σχέδιο έκθεσης και στις τροπολογίες. Άρα μέχρι αύριο ας δούμε κατά πόσο κάτι τέτοιο επαρκεί χρειάζεται ενίσχυση. Αυτά. Νομίζω ότι ε, εξαντλήθηκε και το θέμα επί το παράντος και ο χρόνος. Στις τρεις θα τα ξαναπούμε για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, αν οι συγητές θέλουν να λάβουν το λόγο και θα περάσουμε μετά στις ψηφοφορίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.